Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε το σημείο 4 της μέσης διάταξης με μια μικρή καθυστέρηση, ανταλλαγή απόψεως με τον κύριο, απόψεων με τον κύριο Σέμνεμπι, ο οποίος είναι ειδικός απεσταλμένος για τον Νότιο Κάφκασο, επίσης με τον κύριο Πιέρ Μολέ, ο οποίος είναι ειδικός εκπρόσωπος για την κρίση στη Γεωργία και για τις συνομιλίες της Γενέβης. Έχουμε λοιπόν τη συνολική προβληματική του Καυκάσου και της ε, Γεωργίας. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που μπορώ να καλωσορίσω τους δύο προς και μας και τον κύριο Σέμνεμπι αλλά και τον κύριο Μορέλ. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μορέλ. Όχι, συγγνώμη, τον κύριο Σέμνεμπι θα αρχίσουμε. Σας δίνω το λόγο κύριε Σέμνεμπι. Αλλά προηγουμένως θέλω να επισημάνω ότι θα ακολουθήσει ο συνήθις γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων. Ο κύριος Σέμνεμπι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη χαρά για μένα να είμαι εδώ για τέταρτη φορά ενώπιον της Επιτροπής σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας τον πόλεμο του περασμένου έτους, τον Αύγουστο του 2008, μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας, ήταν ένα καθοριστικό γεγονός στο Νότιο Κάφκασο αυτός ο πόλεμος απίτησε μια αποφασιστική δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι ήρθε στο ύψος των προκλήσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειρηνοποιός δύναμης και ενίσχυσε την εμπλοκή της στην περιοχή αυτή υπογραμμίζοντας και την στρατηγική σημασία του Νοτιού Καυκάσου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συζητήσεις επίση που έλαβαν χώρα για την ε, εταιρική σχέση με το ανατολικά σύνορα της Ευρώπης κάνουν σαφή αυτή τη δέσμευση της Ευρώπης για τα θέματα αυτά παραμένουν ορισμένα ερωτήματα τα οποία πρέπει όμως να απαντήσουμε για τον μέλλον. Θα μπορούσαμε να είχαμε αποτρέψει τον πόλεμο, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Χρειαζόμαστε περισσότερη υποστήριξη στη Γεωργία. Θα πρέπει να είμαστε πιο στεναροί και αυστηροί εναντί τη Γεωργία. Ήμασταν πολύ χαλαροί εναντί τη ε, Ρωσία και τι άλλο θα πρέπει να κάνουμε στην περιοχή. Αυτά σα τα πετάω λιγάκι χήματα, ερωτήματα γιατί είναι χρήσιμο να τα έχετε στο μυαλό σα όταν σκεφτόμαστε για τη μελλοντική πολιτική πρέπει να αναπτύξουμε για την σύνολη περιοχή του Καυκάσου. Οι ευρύτερε τώρα συνέπειε του πολέμου ακόμα δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρω. Είναι γεγονό ότι η δυναμική επέμβαση τη Ρωσία στη Γεωργία έχει οδηγήσει τι χώρε του Νότιου Καυκάσου να καταλάβουν ότι είναι εύθραυστε και τρωτέ, και φυσικά ότι είναι και αλληλεξάρτητε. Η Αρμενία, δύο τρίτα του εμπορίου τη, ακόμα και του εμπορίου τη μέσω τη Ρωσία, περνάει μέσω από τη Γεωργία, είχε μεγάλε διακοπέ προμηθειών σε ενεργειακά προϊόντα υπήρξε απειλή για όλες τις ενεργειακές διαδρομές στην περιοχή του Καυκάσου και σε κάποιες στιγμές διεκόπησαν κιόλας. Αυτή η ιδέα ότι είναι τροτές οι χώρες αυτές λοιπόν του Καυκάσου και επομένως θα πρέπει να αλληλοϊποστηρίζονται, αυτό φάνηκε και από την κοινή προσπάθεια των ε, ε, ειδικών από το Αζερβαϊτζάν και την, ε, που συνεργάστηκαν με του ομόλογου τη Γεωργία για να επισκευάσουν τι υποδομέ έξω από την Τυφλίδα. Υπάρχουν όμω άλλε ε, συγκρούσει οι οποίε υποβόσκουν όπω αυτή που έχει να κάνει με τον Αγκόνο Καραμπάχ μεταξύ Αζερβαϊζάν και Αρμενία και επίση η σχέση τη Αρμενία με την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώ έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο σημαντικό στην υποστήριξη αυτών των προσπαθειών, ιδίω για να ανοίξουν όλα τα σύνορα και οι δύο μεταφορών σε όλη αυτή την περιοχή, κάτι το οποίο θα βελτιώσει πάρα πολύ τη σταθερότητα στον τομέα αυτό στην σύνολη αυτή περιοχή. Τα γεγονότα του Νοτιού Καυκάσου λοιπόν κατέδειξαν σαφώ τη σημασία αυτή τη περιοχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά θέματα στι τρει χώρε που μα ενδιαφέρουν, τα θέματα τη ευκυβερνησίας, των εκλογών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Κράτου δικαίου, όλα αυτά ήταν κατά κάποιο τρόπο άνισα. Ήταν άνισο το ιστορικό στους τομείς αυτούς τα τελευταία χρόνια υπάρχει ο διάλογος φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρεις αυτές κυβερνήσεις των αντιστοίχων χωρών να δημιουργηθεί οικοδόμηση θεσμών και δημιουργία ευκυβερνησίας να προβούν σε ορισμένες ε, συνταγματικές τροποποίησεις οι οποίες θα δώσουν μεγαλύτερη ελευθερία στα μέσα ενημέρωση. Όλα αυτά ήταν ιδιαίτερα επίκαιρα πέρσι, γιατί πέρσι ήταν έτος εκλογών σε όλο τον Νότιο Κάφκασο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά διαδραμάτισε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση των εκλογών στο Νότιο Κάφκασο. Αλλά, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς παρατηρητές θεώρησαν ότι ήταν ε, τίμιες και ε, αδιάβλητες οι εκλογές στις χώρες αυτές, υπάρχουν ακόμα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η κατάσταση οι εκλογές και η ευκυβερνησία των χωρών αυτών. Όλες αυτές οι χώρες λοιπόν έχασαν κάποιες ευκαιρίες να καταδείξουν την πλήρη προσήλωσή τους στη δημοκρατική διακυβέρνηση. Συγχρόνως η έλλειψη βιωσιμότητος ε, των ε, δημοκρατικών θεσμών στις τρεις χώρες παραμένει, παραμένει ένα δημοκρατικό έλλειμμα. Ξεκινώ τώρα με την Αρμενία. Η βία μετά τις εκλογές του 2008 οδήγησε σε 10 νεκρούς και πάνω από 100 ακτιβιστές αντιπολίτευσης που κατέληξαν στις φυλακές. Αυτό κατέδειξε την κατάρρευση της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Το γεγονός ότι συνεχίζονται να κρατούνται και να είναι υπόδικοι ορισμένοι ακτιβιστές αντιπολίτευσης υπογραμμίζει τη σημασία αυτού του πρόβληματος και μας οδηγεί σε ανησυχίες. Εγώ έχω υποστηρίξει την ανάγκη απελευθέρωσης των κρατουμένων την έρευνα σε σχέση με τα γεγονότα του Μαρτίου 2008 να απελευθερωθούν λοιπόν όλοι οι πολιτικοί οι οποίοι έχουν συλλεφθεί και να εφαρμόσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι τα, ε, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για να πω κάτι πιο θετικό, είναι φανερό ότι η αρμενική κυβέρνηση έχει μια, ένα πολύ καλό οικονομικό επιτελείο και πολύ καλή ε, επίδοση στον τομέα αυτό. Έχει προχωρήσει σε φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στον οικονομικό τομέα και έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα για να μεταρρυθμίσει σημαντικά κομμάτια της κρατικής μηχανής, μεταξύ των οποίων την ε, φορολογική και τελωνιακή δίκηση που στο παρελθόν ήταν διαβόητη για την ε, αναποτελεσματικότητά της. Το γεγονό ότι υπήρξε λοιπόν και μια ομάδα εμπειρογνώμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βοήθησε στο ε, εγχείρημα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο τη Γεωργία, η Αρμενία ήταν πάρα πολύ προσεκτική και κράτησε μια στάση ουδετερότητο. Στην αρχή της σύραξης οι αρμενικές αρχές υποστήριξαν τις προσπάθειες εκένωσης από αυτούς, για αυτούς που ήθελαν να φύγουν από τη Γεωργία, διευκόλυνε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γεωργία και βοήθησε τους Ευρωπαίους πολίτες να πάνε και να φύγουν όσοι ήθελαν από την Γεωργία. Ένα αποτέλεσμα της σύγκρουσης Γεωργίας-Ρωσίας ήταν και η προσέγγιση μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας, ιδίως μετά από την προσέλευση του πρόεδρου Γκιουλ στο, σε αγώνα στο Γερεβάν μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας μετά από πρόσκληση του Προέδρου Σαρκισιάν τον Σεπτέμβριο του 2008. Έχουν συνεχιστεί λοιπόν οι προσπάθειες και υπήρξαν και άλλες προ, πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών στις δύο αυτές χώρες μετά από όλα αυτά, ιδίως η πρωτοβουλία για τη συγνώμη σε σχέση με τα γεγονότα του 1915 στην Τουρκία. Για το Αζερβαϊτζάν. Οι αρχές του Αζερβαϊτζάν έχουν και αυτές δείξει το ενδιαφέρον τους να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από την κρίση που έλαβε στη Γεωργία το Αζερβαϊτζάν εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να υπάρξει συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νότιο διάβλο ενέργειας από την Κασπία θάλασσα και έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο να διευκολύνει τις επαφές μεταξύ του Ορμενιστάν και Τουρκίας για τους ενεργειακούς διάβλους και εξακολουθεί να είναι προσιλωμένο στην ιδέα του διάβλου αυτού που θα διασχίζει την Κασπία για να εξασφαλίσει και τη βιωσιμότητα του Ναμπούκου μετά από τον πόλεμο της Γεωργίας, μία από τις σημαντικότερες συμβολές του Αζερμπαϊτζάν στη σταθεροποίηση της περιοχής ήταν η δέσμευση να συνεχίσει να δίνει φυσικό αέριο στη Γεωργία. Οι προεδρικές εκλογές του Αζερμπαϊτζάν που μποϊκοταρίστηκαν από ένα μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης μπορούν να θεωρηθούν ότι ήταν καλά οργανωμένες και τακτικές αλλά σε τελική ανάλυση δεν καλύπτουν τα πρότυπα του δημοκρατικού πλουραλισμού. Η απόφαση στις 18 Δεκεμβρίου του Κοινοβουλίου του Αζερμπαϊτσάν να καταργήσει το όριο των δύο θητιών για τον πρόεδρο της χώρας μπορεί να μειώσουν τις δυνατότητες πολιτικής πολυμορφίας στο μέλλον. για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα μέσα ενημέρωση. Είναι ανάμεικτη η κατάσταση του Αζερμπαϊτσάν. Ορισμένε προσπάθειε για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατεβλήθησαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, όπω παραδείγματο χάρη η εφαρμογή της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, την ε, απελευθέρωση κρατουμένων δημοσιογράφων, την εξέταση κάποιων εκθέσεων για βία από την πλευρά του στρατού κτλ. Αλλά στις 30 Δεκεμβρίου παρόλα αυτά το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο δεν ανανέωσε την άδεια ορισμένων εταιριών που είχαν ξένους ιδιοκτήτες, κάτι το οποίο έχει επικριθεί από τη διεθνή κοινότητα μεταξύ των οποίων και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πρόσκομα για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης για το Άνω Καραμπάχ. Δεν θα πω πολλά πράγματα, αλλά υπήρξαν κάποιες θετικές εξελίξεις μετά από τον πόλεμο της Γεωργίας. Ιδίως στις 2 Νοεμβρίου η Ρωσία έκανε μια δήλωση βάσει της οποίας για πρώτη φορά οι, τα δύο μπλεκόμενα μέλη ε, αποδέχονται τις αρχές της Μαδρίτης που είχαν διατυπωθεί για αυτή τη σύραξη. Παρά όλα αυτά η κατάσταση παραμένει αντιφατική. Υπήρξαν δηλώσει από τη μεριά του Αζερμπαϊτζάν που φαίνεται ότι δείχνουν ότι δεν είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους και φυσικά επικρίνουν την ηγεσία της Αρμενίας και έχουμε και ορισμένες παραβιάσεις και από τις δύο πλευρές της συμφωνίας ε, κατάπαυσης του πυρός και απεμπλοκής. Γεωργία τέλος. Στην Γεωργία η εσωτερική πολιτική, οικονομική και κατάσταση ασφαλείας. Είναι σταθερή αυτή τη στιγμή, αλλά είναι αρκετά εύθραυστη αυτή η σταθερότητα. Η οικονομική κρίση, η οποία έχει επηρεάσει πολύ σοβαρά την Γεωργία, λόγω του πολέμου του 2008 και της επερχόμενης χρηματοοικονομικής κρίσης ανάγκασε την κυβέρνηση Γεωργίας να εστιάσει την προσοχή της σε κοινωνικο-οικονομικά θέματα και όχι θέματα εδαφικά. Αυτό όμως θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον, θα μπορούσε ραγδαίως και άρδιν να αλλάξει αν επιδεινωθεί η κατάσταση, γι' αυτό θα πρέπει να παραμένουμε άγρυπνοι σε σχέση με την κατάσταση αυτή. Η Γεωργία είχε πολλές εκλογές, και κοινοβουλευτικές, περιφερειακές και προεδρικές εκλογές πέρυσι το 2008. Δεν υπήρξε συνένεση σε σχέση με το πώς έπρεπε να διαργηθούν αυτές οι εκλογές και έγιναν με ένα ιδιαίτερα πεπολωμένο τρόπο σε ένα απολωμένο πολιτικό κλίμα. Σε ό,τι αφορά την Νότια Οσετία και την Απχαζία, ο Πιέρ Μορέλ θα αναφερθεί στο θέμα αυτό, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Εγώ θέλω να πω απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Αποστολή Παρακολούθησης έχει διαδραματίσει ένα σημαντικό σταθεροποιητικό ρόλο και το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στις ε, υποαπόσχεις αυτές τις περιοχές δεν επέτρεψε στην ε, αποστολή μας να εκπληρώσει πλήρως την εντολή μας, εντολή τους. Για να μπορέσουμε λοιπόν Έχουμε και άλλα θέματα φυσικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το θέμα των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, IDPs στα αγγλικά, το οποίο θα αναφέρει ο Πιέρ Μορέλ για το μέλλον της διεθνούς παρουσίας στην περιοχή του Κάσου και όπου η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία από τις τρεις αποστολές αυτή τη στιγμή είναι η μόνη αποστολή που έχει μια εντολή που ξεπερνάει το Φεβρουάριο του 2009. Το θέμα λοιπόν των εντολών αυτών των αποστολών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παραμείνει ή στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μας. Μαζί με άλλους συνομιλητές εγώ ζήτησα από τις γεωργιανές αρχές να διερευνήσουν τα γεγονότα του 2008, του Αυγούστου 2008. Αυτό έχει γίνει από μια κοινοβουλευτική επιτροπή που ήταν μια πρωτοφανή τέτοια επιτροπή για τη γεωργία και επίσης όπως ζήτησε και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητούσε μια διεθνή έρευνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε τη δική της έρευνα για τα γεγονότα του Αυγούστου 2008 η οποία γίνεται, όπως σας είπα, με ένα ανεξάρτητο τρόπο από την Κομισιόν και θα παρουσιαστεί τα πορίσματά της μέχρι τον Ιούλιο του 2009. Είναι πολλέ λοιπόν οι δραστηριότητε, είναι πολλά τα σχέδια τα οποία εκτιλήσονται στον Κάφκασο και είχαμε πολλά τέτοια σχέδια στις υποαπόσχεση περιοχές πριν από τον πόλεμο του 2008. Πολλές από αυτές θεώρησαν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν τα κοινά του συμφέροντα και να έχουν ένα μια καλύτερη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά από αυτά τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη μπορούν να συνεχιστούν χωρί να υποσκάψουν την υποστήριξη για την εδαφική ασφάλεια και ακαιρεότητα τη Γεωργία και από την άποψη αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει και μέσω εμού να είναι σε επαφή με τη Γεωργία για την ομοθεσία σε ό,τι αφορά τα κατεχόμενα εδάφη και με τον τρόπο με τον οποίο τα σχέδια αυτά μπορούν να ευθυγραμμιστούν με την νομοθεσία τη Γεωργία. Εν κατά κλείδι, ο πόλεμος στη Γεωργία κατέδειξε ότι τα προβλήματα του Καυκάσου είναι θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα τα προβλήματα αυτά. Όλα αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν επίσης να αποχωριστούν από τις σχέσεις μας με τις δύο μεγάλες δυνάμεις και εταίρους μας σε αυτήν την περιοχή, την Ρωσία και την Τουρκία. Όσο προβληματική μπορεί να είναι και η σχέση μας με τη Ρωσία τον Αύγουστο, δεν μπορούμε να την βγάλουμε το παιχνίδι. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες για μια συνολική αντιμετώπιση, οι πρωτοβουλίες για μια εταιρική σχέση, οι συναντήσεις υψηλού επίπεδου που θα λάβουν χώρα τους επόμενους μήνες για να προωθήσουμε την ε, παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ε, νότιο διάβλο ενέργειας, καθώς και οι διαπραγματεύσεις που κάνουμε σε σχέση με τις διάφορες συνθήκες με τη Ρωσία και οι πολυσχηδείς και πολυεδρικές μας σχέσεις με την Τουρκία και εδώ, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ταυτοποιηθεί ως ε, εταίρος την πρωτοβουλία της Τουρκίας για μια περιφερειακή πλατφόρμα για τον Νότιο Κάφκασο. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε πολύ φαΐ στο πιάτο μας, πολλά πράγματα να κάνουμε και ελπίζω μέχρι την επόμενη μου παρουσία να υπάρχουν στην Επιτροπή σας, να υπάρχουν και νέα τα οποία μπορώ να σας αναφέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε και τώρα δίνουμε το λόγο στον κύριο Μορέλ, ο οποίος θα μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη Γεωργία. Κύριε Πρόεδρε, <clears throat> χαίρομαι που παίρνω το λόγο ως ε, ειδικό αντιπρόσωπος για την κρίση στη Γεωργία. Πολλές φορές ε, έχω πάρει το λόγο εδώ για την αποστολή μου στην Κεντρική Ασία γενικά, η οποία συνεχίζεται, αλλά η κρίση της Γεωργίας είναι μία θα ονόμαζα ad hoc κρίση και γι' αυτό συνεργάζομαι ε, με τον κύριο Σένεμπι προσπαθώντας να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε τις τελευταίους ε, μήνες. Προσπαθούμε λοιπόν να συνεργαστούμε και με την αποστολή παρατήρησης τον πρέσβη Χάμπερ και των ε, στρατηγό Ζαμπέρ και συνεργαζόμαστε φυσικά και με τις ε, διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών στην περιοχή. Επαναλαμβάνω ότι η εντολή μου καλύπτει την κρίση στην Γεωργία ως έχει σήμερα. Πρόκειται για μια αποστολή επαναλαμβάνω ad hoc η οποία έχει σαν στόχο να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια την οποία κάνει και να σας εξηγήσω γιατί. Πρώτον, αυτό το κάνουμε μέσω μιας γενικής αξιολόγησης της κατάστασης και δεύτερον μέσω των προσπαθειών των συνομιλιών της Γενέβης. Πρέπει να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω ότι η σύγκρουση στη Γεωργία είναι μια παλαιά σύγκρουση. Η ιστορία της ολοκλήρωσης για δύο αιώνες και της συμπερίληψης της Γεωργίας στην Ρωσική Αυτοκρατορία καταρχάς και στη Σοβιετία ε, κατά δεύτερον είναι κάτι το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι γνωστό και τεκμηριωμένο. Ε, ξαναβρήκε την εθνική ταυτότητα σαν πρώτο χριστιανικό βασίλειο με την Αρμενία το οποίο διαδέχτηκε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μια ανεξαρτησία όμως την οποία έχασε ε, μετά από λίγο καιρό το 1921 Υπάρχει δηλαδή πέραν της μακράς διάρκειας στην ιστορία και μια σύγχρονη σχετικά εικόνα για την ανεξαρτησία της Γεωργίας. Θυμηθείτε τον Στάλιν, θυμηθείτε επίσης ε, αυτά τα οποία έκανε ο Μπέρια στην Απχαζία, ο οποίος Μπέρια ήταν Γεωργιανός και όλα αυτά έχουν θεμέλια ιστορικά λοιπόν τα οποία είναι βαθύτατα και βαρύτατα Ίσως η σύγκρουση αυτή να οφείλεται τελικά και στις συνέπειες της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης μετά από εθνικιστικές κινητοποιήσεις του Προέδρου Γκαμσακουρία, παλιού αντιστασιακού εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, αυτός ο εμφύλιος πόλεμος οδήγησε σε 20.000 νεκρούς. Ήταν μια τραγωδία η οποία δεν ανοιχνεύτηκε ποτέ επί της ουσίας και όλα αυτά συνθέτουν θα έλεγα τον ιστό πάνω στον οποίο προσπαθεί να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαν δημιουργηθεί δύο μηχανισμοί επαφής, διαχείρισης, ελέγχου της μετεμφυλιακής κατάστασης. Καταρχάς, το JCC, η Μικτή Επιτροπή για την Νότια Οσετία επί τη βάση της Συμφωνίας του Σότσι του 1991. Υπάρχει επίσης και η ομάδα φίλων της Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών μετά τη συμφωνία του 1994 στη Μόσχα. Και υπάρχει και η Μονίκη, αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Εθνών στην ίδια τη Γεωργία. Ένα σύστημα το οποίο λειτουργούσε, με κάποια εμπόδια βέβαια αλλά σιγά σιγά οι διαπραγματεύσεις οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο και με τη σειρά του το αδιέξοδο αυτό προκάλεσε τις συγκρούσεις στο θέατρο των επιχειρήσεων. Δεν θα επανέλθω τώρα στην διαδοχή των γεγονότων του Ιουλίου και του Αυγούστου. Αυτά σας τα υπεθύμησε και ο Πέτες Ένμπι. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυρία Ταλιαβίνη αλλά αυτό που έχει σημασία για μας όλους εδώ είναι ότι η προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την περιοχή αυτή είναι απόλυτα δικαιολογημένη γιατί είναι η πρώτη διεθνής κρίση της οποίας μάλλον επιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ότι το θελήσαμε αυτό από μόνοι μας ή το επιδιώξαμε. Οι συνθήκες μας οδήγησαν θα έλεγα. Θυμίζω ότι πέντε μήνες μετά το τέλος της κρίσης της οξυμένης νομίζω καταλήγουμε σε τρία πρώτα συμπεράσματα. Πώς έγινε αυτό το οποίο έγινε. Τρεις ήταν οι αιτίες. Πρώτον, υπήρξε μια επαναδραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν δυνατότητες πρωτοβουλίας, τις χρησιμοποίησε η Γαλλική Προεδρία, έπαιξε ένα κυρίαρχο ρόλο αν εμφυμίστε από τις 8 μέχρι τις 12 Αυγούστου υπήρξαν πάρα πολλά πηγενέλα από το Παρίσι στην περιοχή ε, και επίσης ε, προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε και το Συμβούλιο Ασφαλείας αλλά είχε μπλοκαριστεί εντελώς. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τον ΟΑΣΕ και εκεί δυστυχώς είχαν μπλοκαριστεί τα πράγματα. οι σχέσεις της γεωργίας, μιας νέας γεωργίας η οποία είναι κοντά στις Ηνωμένε Πολιτείε πλέον είναι κάτι το οποίο δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στη διαχείριση των προβλημάτων της περιοχής. Γι' αυτό λοιπόν η ευθύνη στην ουσία περιέπεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω της δραστηριότητας του Προέδρου Σαρκοζή εμείς επιμείναμε για την εφαρμογή της συμπληρωματικής συμφωνίας της 8 η Σεπτεμβρίου. Υπήρξαν επανειλημμένες συναντήσεις ανάμεσα στον πρόεδρο Μπαρόσο και στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, ανάμεσα στον κύριο Σολάνα και εκπροσώπους των εμπλεκομένων χωρών η δημιουργία μιας Επιτροπής Ελέγχου και Παρατήρησης. Αρχές Οκτωβρίου ξεκίνησε η επίσημη αποστολή. 10 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η απόσυρση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από την Απχαζία και τη Γεωργία και στις 13 Οκτωβρίου ξεκίνησε μια διάσκεψη στη Γενέβη και στις Βρυξέλλες λίγο αργότερα μια συνάντηση των δωρητριών χωρών. Όλα αυτά τα επιδιώξαμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και ρυθμό. Δεύτερο μάθημα, κινητοποιήσαμε όλα τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας, δηλαδή καταρχάς την Επιτροπή Παρατήρησης και Ελέγχου, ένα ε, μήνα λειτουργούσε, ιδρύσαμε όμως σε άλλες τρεις περιοχές ε, γραφεία, συμμετέχουν 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε μια τεράστια προσπάθεια από πλευρά των δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν παρούσες στη Γεωργία, που είναι παρούσες, κινητοποιήσαμε τους μέγιστους δυνατούς πόρους για μια αποστολή πάρα πολύ δύσκολη, χωρίς όπλα και αυτό ήταν σκεμμένο βέβαια, σε μια περιοχή παρόλα αυτά επικίνδυνη και καταφέραμε να συλλέξουμε την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε ε, τι συμβαίνει ε, σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι συζητήσεις που γίνονται ακούγονται η ε, Πρίστινα, το Σεράγεβο, η Γάζα, Δηλαδή ακούγονται καταστάσεις εντελώς διαφορετικές οι οποίες γίνονται μερικές φορές αντικείμενο αναφοράς από τους συνομιλητές μας. Όλα αυτά προσπαθήσαμε όμως να τα αντιμετωπίσουμε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ήρθαμε σε επαφή με το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Γεωργίας, συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Άμυνας της Ιδίας Χώρας, Ατέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, οι προσπάθειες τις οποίες κάναμε πήραν και διαφορετική μορφή. Κάναμε 1.400 επί τούτου αποστολές από τότε μέχρι σήμερα από τις οποίες 250 τη νύχτα. 250 νυχτερινές αποστολές παρατήρησης. Μόνο εμείς κάνουμε νυχτερινές αποστολές παρατήρησης. Όπως είπα κινητοποιήσαμε τα πάντα, τη γραμματεία του Συμβουλίου, τον Πέτερ Σένεμπι, τον ειδικό εκπρόσωπο δηλαδή για την κρίση στη Γεωργία. Από τις 15 Οκτωβρίου και μετά προετοιμάσαμε τη συνάντηση της Γενέβης, ιδιαίτερα την εβδομάδα την προπαρασκευαστική της ε, συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών διάσκεψη των δωρητριών στις 22 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες που επέτρεψε μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την αιγίδα των Μπαρόζο και Φεραίρο Μπάλνερ να κινητοποιήσουμε 5.700.000 δολάρια σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία αλλά και με συγκεκριμένους πολιτικούς όρους βοήθεια πολιτική προς τον γεωργιανό πληθυσμό με διαφάνεια και έλεγχο και με υποχρέωση του υπόλογου κάθε φορά αυτού ο οποίος παραλαμβάνει και διανέμει τη βοήθεια. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι η συνοχή την οποία επέδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θα πρέπει να αναφερθώ στις πρώτες έκτακτες συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών και στο έκτακτο συμβούλιο της 1ης Σεπτεμβρίου. Το συμβούλιο αυτό ξεκαθάρισε μια στοχευμένη γραμμή απέναντι στην κρίση, μια σαφέστατη ε, προϋπόθεση την αναγνώριση των προσπαθειών αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μόσχα, ένα μήνυμα σχετικά σταθμισμένο αλλά και σκληρό προς τη Μόσχα, την καλέσαμε να υπολογίσει το βάρος των ενεργειών της, Νομίζω ότι στείλαμε το πολιτικό μήνυμα το οποίο έπρεπε, το δέον πολιτικό μήνυμα, ένα ισχυρό και ισορροπημένο, το οποίο θα έλεγα δείχνει ότι υπάρχει μια συνοχή των θέσεων στις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν υπάρχουν διαιρέσεις και γι' αυτό καταλήξαμε σε μια συμβιβαστική με λύση, δυναμικά όμως συμβιβαστική λύση η οποία στηρίζει τις θέσεις μας. Παράλληλα, προσπαθήσαμε να σεβεστούμε όλες τις χρονικές προθεσμίες. Η συγκέντρωση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών τοποθέτησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά πρωτοπόρα στη διαχείριση της κρίσης και όχι ένας απλός σε εισαγωγικά συνεισφορέας όπως το παρελθόν. Αυτό είναι το μάθημα που πήραμε από τη Γεωργιανή κρίση. Και αυτό είναι και μια υποχρέωση βέβαια η οποία δημιουργείται για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον Βλέπουμε ότι όλα αυτά βασίζονται και στις συζητήσεις της Γενέβης και όλα αυτά δείχνουν την πολιτική δουλειά που πρέπει να γίνει, ιδιαίτερα στη Γενέβη. Οι αρχές ήταν δύσκολες λοιπόν, δεν υπήρχαν προηγούμενα το σύστημα ε, των διπλωματικών σχέσεων ε, με τη Ρωσία διεκόπηθα, θα έλεγα μετά από πρωτοβουλία της Γεωργίας και διεκόπησαν επίσης ε, και οι συνθήκες του Σότσι οι οποίες διαχειριζόντουσαν άλλοτε καλά και άλλοτε άσχημα τα προβλήματα από το 1992 και μετά. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο πολιτικών επαφών επί τη βάση του άρθρου 6 της Παλαιάς Συμφωνίας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Έγιναν επίσης και κάποια μικρά βήματα στην εφαρμογή της συμφωνίας της 8 η Σεπτεμβρίου. Δύο μήνες μετά τον πόλεμο υπάρχει πάντα αμοιβαία απόρριψη ανάμεσα στη Γεωργία και τη Ρωσία σε εξαιρετικά σκληρές προϋποθέσεις και από πλευράς ρωσικής και από πλευράς ε, ε, γεωργιανής είτε στο Τσιγκφάλι είτε στο Σουχούμι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γραμματεία του Συμβουλίου ε, στην ουσία συμμετέχουν στις συζητήσεις της Γενέβης μαζί με τον ΟΑΣΕ και τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς στείλαμε, επαναλαμβάνω, παρατηρητές μας εκεί. Υπήρχαν και παρατηρητές του ΟΑΣΕ στην Οσετία του Νότου, αλλά υπήρχαν και κινήσεις στρατευμάτων στην Αμπχαζία όπου εκεί δεν ξέσπασε πόλεμος, δεν ξέσπασαν συγκρούσεις. Υπήρχε όμως παρουσία και της και εκεί των Ηνωμένων Εθνών οπότε και οι τρεις μαζί προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε. Ο ΑΣΕ, ο ΙΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενότητα παρουσίας και δράσης στον χρόνο και στον τόπο. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε λοιπόν την επιστροφή στην ε, εξομαλυμένη θα έλεγα κατάσταση αυτό αρχίσαμε να το πετυχαίνουμε συμβολικά στις 14 Οκτωβρίου το βράδυ με ένα δείπνο στη Γενέβη πριν από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι επίσημες διαπραγματεύσεις. Το δείπνο αυτό ήταν ένα δείπνο εργασίας, ακούστηκαν συγκεκριμένες θέσεις και προς τον τύπο μετά το δείπνο αυτό από τη Γαλλική Προεδρία, από τα ευρωπαϊκά όργανα, από τον κύριο Κούσνερ, από τον κύριο Σολάνας, από την κυρία Βάλνερ, από τον Μπαν Κι Μουν και από τον κύριο Γκουτιέρες, επίτροπο ανώτατο Ήπατο για, τα Ηνωμένα, ε, για τους ε, πρόσφυγες, τον κύριο Στούμπ, εκπρόσωπο ε, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης, μάλλον του, του Συμβουλίου Υπουργών του ΟΑΣΕ και επίσης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ πάντα. Υπήρξε δηλαδή μία συντονισμένη προσπάθεια των τριών θεσμικών οργάνων για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασής τους... στο πλαίσιο το οποίο έχω ήδη περιγράψει. Μια άλλη δυσκολία είναι το θέμα της μορφής αυτών των διαπραγματεύσεων. Στην ουσία η Ρωσία ήθελε να διαχειριστεί σε διμερές επίπεδο με τον Σαρκοζή τη Γαλλική Δημοκρατία δηλαδή τις συζητήσεις στη Γενέβη. Βέβαια μιας και οι ρωσικές δυνάμεις έπρεπε να αποχωρήσουν δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τις διαπραγματεύσεις αυτές με τέτοιο τρόπο. Υπήρξαν λοιπόν εξ αρχής τακτικές και συμβολικές αντιρρήσεις για την Αμερικανική σαν παράδειγμα παρουσία στη Γενέβη, κάτι το οποίο δεν ήταν και εύκολο να ξεπεραστεί. Ε, το θέμα της ε, αναγνώρισης ή μη αναγνώρισης της ταυτότητας της Γεωργίας όχι από τη Ρωσία αλλά από όλους τους άλλους συμμετέχοντες στη Γενέβη δημιουργήσαμε δηλαδή μια δομή διαπραγματευτική περίπλοκη μορφής 6 συν 2 τρεις συμπρόεδροι Ρωσία, Γεωργία, Ηνωμένε Πολιτείε συν δύο εμπλεκόμενες ε, πλευρές στην ουσία δηλαδή δημιουργήθηκε μια ολομέλεια ανάμεσα σε κράτη τα οποία έχουν διεθνή ταυτότητα και δυνατότητα διεθνούς παρουσίας αλλά και συμμετοχή όλων των υπολείπων ενδιαφερομένων με συγκεκριμένες μορφές δυνατότητας παρέμβασης τις οποίες ρυθμίσαμε λεπτομερώς πλέον αλλά με τον χρόνο. Μια ομάδα εργασίας η οποία προεβλέπεται από τη συμφωνία της 12ης Αυγούστου αλλά και αυτήν της 8ης Σεπτεμβρίου, ομάδα σταθεροποίησης της περιοχής πρώτον και η δεύτερη ομάδα, ομάδα διαχείρισης των προβλημάτων των εκτοπιστέντων και των προσφύγων. Ξέρετε ότι για τη Ρωσία αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα γιατί πρόσφυγας θεωρείται αυτός που πάει σε μια άλλη χώρα. Αλλά οι κάτοικοι της Αμχαζίας όταν περνούν στην υπόλοιπη Γεωργία θεωρούνται εκτοπιστέντες για τους Γεωργιανούς και όχι πρόσφυγες. Βλέπετε ότι ακόμα και οι μικρές λέξεις μερικές φορές γίνονται αιτία όρθωσης ε, μεγάλου εμποδίου. Μεγάλη σημασία λοιπόν έχουν οι επαφές τις οποίες έχουμε επιτόπου όταν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά. Απαιτείται χρόνος λοιπόν να ξεκινήσουμε, παρόλα αυτά ξεκινήσαμε, ε, διανύσαμε κάποια στάδια. Η Γενέβη 1, 15 Οκτωβρίου ξεκίνησε γέρος στα πλαίσια διεθνούς έντασης και πίεσης μπορέσαμε να υιοθετήσουμε κάποιες κανόνες λειτουργίας, κάποιους κανόνες λειτουργίας, υπήρξαν κάποια αμοιβαία μποϊκοτάζ σε ορισμένες συζητήσεις ανάμεσα στους Ρώσους και τους Γεωργιανούς, Παρόλα αυτά έγιναν οι παράλληλες συζητήσεις, έγιναν οι εκ του διαπραγματεύσεις, τα proximity talks και νομίζω ότι τελικά κάποια στιγμή μπορέσαμε να αρχίσουμε να επικοινωνούμε και οι Ρώσοι με τους Γεωργιανούς. Βρήκαμε μετά από αυτή τη δύσκολη εκκίνηση μια δεύτερη ημερομηνία για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Όλοι εξεφράστησαν και όλοι αποφάσισαν να συναντηθούν σε μια ευθετότερη χρονική στιγμή. Φτάνουμε λοιπόν στην Γενέβη 2 θα την ονομάσω. Είχαμε προετοιμαστεί σωστά, είχαμε προπαρασκευαστεί σε σχέση με τον εντοπισμό των θυμάτων. 18 του μηνός το βράδυ ξεκινήσαμε με ανεπίσημο δείπνο, όλοι ήταν παρόντες εκεί χωρίς εξαιρέσεις. Άρχισαν να συνεδριάζουν οι δύο ομάδες εργασίας τις οποίες σας έχω περιγράψει εκ παραλίλου. Επαναλαμβάνω η ομάδα εργασίας 1 ασχολείται με θέματα ασφαλείας συμπροεδρεύεται από τους τρεις συμπροέδρους γιατί τα θέματα ασφαλείας εμπλέκουν θα έλεγα όλες τις ε, δυνατότητες ενδράσεις που έχει ο ΑΣΕ, τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ η ομάδα εργασίας 2 συμπροεδρεύεται από ένα εκπρόσωπο τον κύριο Βιγκό εκπρόσωπο της ΡΕΛΕΞ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από έναν εκπρόσωπο της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες τον κύριο Γένς από τη Γενέβη. Μπορέσαμε λοιπόν να εντοπίσουμε τα θέματα επί των οποίων έπρεπε να εργαστούμε για να ξεκινήσουμε και τη Γενέβη 3 από τις 10 Δεκεμβρίου. Εκεί εργαστήκαμε παράλληλα 9 ώρες, εκ παραλλήλου 9 ώρες το Δεκέμβριο η ομάδα 1 συγκέντρωσε τις προσπάθειές της στους μηχανισμούς πρόληψης των ε, αρνητικών συμβάντων, υπήρξαν συμφωνίες σε πολλά θέματα, υπήρξαν κάποιες τελευταίες επιφυλάξεις για το καθεστώς των περιοχών από τις δύο πλευρές, υπήρξε μια θα έλεγα αναβολή της τελικής συμφωνίας, παρόλα αυτά ε, αισθανθήκαμε ότι όλοι θέλουν να καταλήξουμε κάπου σε διαδικασίες πρόληψης ε, των αρνητικών συμβάντων. Μιλήσαμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ε, δυνατότητες ελέγχου, κοινέ επισκέψεις των παρατηρητών και των δυνάμεων ελέγχου της κατάστασης. Η ομάδα 2 ασχολήθηκε με την ανθρωπιστική βοήθεια, την εξιολόγηση των της, του βαθμού δυσκολίας στην οποία βρίσκονται οι πρόσφυγες και οι εκτοπιστέντες. Συνεχίζονται, εν πάση περιπτώσει, οι διαπραγματεύσεις της Γενέβης και οι δύο εμπλεκόμενες δυνάμεις, χώρες μάλλον, βρίσκουν ενδιαφέρον στις επαφές αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν λοιπόν οι επαφές αυτές, είναι κάτι το μακροπρόθεσμο, έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά που είναι μάλλον σωστή δουλειά. Η Ρωσία πάει σταδιακά και βραχυπρόθεσμα. Δεν θέλει να υπάρξει μια δεύτερη διαδικασία του Μίνσκ όπως είπε ο Σένεμπι ούτε και εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν μπορούμε να σαλαμοποιήσουμε την κρίση εμείς μετά από λίγους μήνες, μια κρίση η οποία έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Πήραμε πρωτοβουλίες λοιπόν και τις πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να τις ολοκληρώσουμε βασιζόμενοι στα συγκεκριμένα προβλήματα αλλά με μια ξεκάθαρη πολιτική. Στη Γενέβη θα πρέπει να λάβουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με τον ΟΗΕ και με τον ΟΑΣΕ ε, προσεκτικά και θα πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε τον ρόλο τον οποίο έχουμε ξεκινήσει. Οι επαφές της Γενέβης δεν είναι επίσημη διαπραγμάτευση, δεν είναι ούτε καν μια τυπική διάσκεψη. Είναι μια άτυπη πολιτική διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει και κατά τη διάρκεια των επομένων μηνών μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν διαρθρωμένο μηχανισμό ελέγχου της γεωργιανής κρίσης. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας κύριε Πρεσβευτά. Για το γεγονός επίσης σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας λίγο πριν φύγετε για τα Ηνωμένα Έθνη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σύντομοι γιατί στις 4 και 10 πρέπει να φύγετε για το αεροδρόμιο. Αυτό είναι το μάξιμου νομίζω που μπορώ να εξασφαλίσω από εσά κύριε Μορέλ. Προτείνω λοιπόν ο πρώτος γύρος ερωτήσεων να αφορά το τμήμα του κυρίου Μορέλ. Και πρωτού δώσω το λόγο σε αυτούς που θέλουν να λάβουν το λόγο, σας ζητώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι πρώτον, γιατί στις 4 και 10 όπως είπα σε 13 λεπτά πρέπει να φύγει ο κύριος Μορέλ και θέλω να χαιρετήσω τα νέα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Κύριτα από τη Ρουμανία που αντικαθιστά. Που αντικαθιστά την κυρία Αναστάζε. Παίρναμε τώρα στις ερωτήσεις που θέλουν να θέσουν τα μέλη μας. Σας παρακαλώ να είστε όσο δυνατόν λακωνικότεροι και εστιάστε παρακαλώ στο τμήμα που έχει να κάνει με τη γεωργία η κυρία Ισλέρ Μπεγκέν, που είναι η επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τον Νότιο Κάφκασο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μορέλ για την παρουσίασή σας. Δεν συμμερίζομαι απόλυτα αυτά τα οποία είπατε, γιατί στην αρχή δεν αναφέρατε κάτι το γεγονός ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολλούς μήνες ήμασταν επάγρυπνοι και είχαμε προειδοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε μια πολιτική πρόληψης που κατά την άποψή μας ή ορισμένο από μας θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την κλιμάκωση στη Γεωργία και τον πόλεμο ο οποίος ε, εξέσπασε στη Γεωργία. Σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώσουμε ότι έχουν αλλάξει οι συντεταγμένες. Πριν από τη σύγκρουση είχαμε απλώς μια διοικητική οριοθετική γραμμή μεταξύ της Νότιας Οσετίας και της Γεωργίας. Τώρα ουσιαστικά πρέπει να μιλήσουμε για σύνορα εφόσον είναι αδιαπέραστη αυτή η γραμμή, εφόσον κανείς δεν μπορεί να περάσει από τη μία περιοχή στην άλλη, <coughs> δεν μπορούμε να μιλήσουμε παρά μόνο για σύνορα. Μιλάμε λοιπόν ακόμα για εδαφική ακαιρεότητα της Γεωργίας. Τι θα πει εδαφική ακαιρεότητα όταν εμείς ως Ευρωπαίοι μιλάμε για το σεβασμό της εδαφικής ακαιρεότητας της γεωργίας. Έχετε κάποια ελπίδα ώστε κάποτε θα υπάρξει ένα συνολικό καθεστώς για αυτές τις περιοχές. Γιατί σήμερα έχουμε την αποστολή αυτή, δεν ξέρω αν ο ΙΕ θα μπορέσει να γυρίσει στην περιοχή. Η Ρωσία έθεσε βέτο στην παρουσία της αντιπροσωπείας της ΟΑΣΕ. Με έχουμε μονάχα τους παρατηρητές Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτοί είναι παρακολουθητικές και δεν μπορούν να παρέμβουν. Ευχαριστώ κύριος Κασουλίδης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μορέλ ορισμένα συγκεκριμένα θέματα. Καταρχήν, σε σχέση με τον εντυπωσιακό ρόλο, όπως υπογραμμίζω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο μας παριέγραψε, το ρόλο του πρόεδρου Σαρκουζή και της Γαλακής Προεδρίας. Αλλά εδώ αναρωτιέμαι, οι Ηνωμένε Πολιτείε που δεν θέλησαν να διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο στην περιοχή αυτή, υπήρξε κάποιος λόγος συγκεκριμένος για τον οποίο άφησαν περιθώριο και ένα κενό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να το καλύψει. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι, μιλάμε για τις λεγόμενες παγωμένες σειράξεις όπως την Απχαζία και την Νότια Οσετία. Αλλά δεν είναι παγωμένες γιατί άμα τίκονται αυτές οι σειράξεις έχουμε πολέμους όπως αυτός του τελευταίου καλοκαιριού. Μήπως το θέμα αυτών των ε, παγωμένων σειράξεων απλώς καθησυχάζει την παγκόσμια κοινότητα και την αποτρέπει από το να έχει μια συγκεκριμένη δράση για να αποτρέψει τέτοιες συγκρούσεις. Ευχαριστώ. Thank you. Um, what is your assessment on the recommendation? Ποιε είναι οι δικοί σα ε, οι εκτιμήσεις σχετικά με τις ίσες κομισιόν για την, ε, ανατολική, για την συνεργασία προς Ανατολάς. Και επίσης στην ε, πλατφόρμα του Καυκάσου θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα να βελτιωθούν οι σχέσεις με τη Γεωργία και με άλλες χώρες του Νοτιού Καυκάσου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω εσείς ε, θεωρείτε ότι οι προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται σε δύο συμφωνίες που υπογράφηκαν τον Οκτώβρη ε, καλύπτονται αυτές. Και έχω κατά νου τρία πράγματα κυρίες. Πρώτον, το μελλοντικό καθεστώς της Απχαζίας και της Νότιας Οσετίας που υποτίθεται ότι θα συζητήσουμε. Αυτό όμως έχει ήδη κατά κάποιον τρόπο προαποφαστεί από τη Ρωσία. Εσείς τι πιστεύετε από αυτού. Δεύτερον, ε, υπάρχει το θέμα της απόσυρσης ε, των ε, στρατευμάτων στις θέσεις που υπήρχαν πριν από τη σύραξη και το θέμα αυτό δεν έχει λυθεί ακόμα. Και τέλος, ε, η πρόσβαση των παρατηρητών. Οι δικοί μας οι παρατηρητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα τμήματα της Νότιας Οσετίας, ακόμα και σε εκείνα που κατοικούνται αποκλειστικά και μόνο από Γεωργιανούς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, χωρίς μικρόφωνο βέβαια. Ο μιλητής εξακολουθεί να ευχαριστεί χωρίς μικρόφωνο. Le Μικρόφωνο παρακαλώ επισημαίνει ο Πρόεδρος. Συγγνώμη. Κύριε Πρέσβη, κατανοώ ότι είναι σαφής ο στόχος σας ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, επαναφορά της ειρήνης, της μόνιμης ειρήνης στον Κάφκασο και όλοι συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη. Μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες όμως που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι δύσκολη η απάντηση στο ερώτημα αυτό του πώς θα επιτευχθεί γιατί πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και δεν θα είναι εύκολες. Αλλά με ποιο σημείο εκκίνησης κύριε Πρέσβη εσείς δεσμεύεστε στις διαπραγματεύσεις αυτές. Τι θέλουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θέλουμε να προτείνουμε, τι θέλουμε να επιβάλλουμε, τι θέλουμε να εξασφαλίσουμε από αυτέ τι διαπραγματεύσεις. Μπορούμε να δούμε τι θέλουν οι Ρώσοι, οι Απχάσοι και οι Γεωργιανοί. Αλλά επειδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση σύγκρουσης που είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί, υπάρχει από τη δική μας πλευρά ένα σενάριο, μια ιδέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι είναι το πρακτέον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ανδρέας Νταφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον η Γεωργία εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Γεωργία εξακολουθεί να πιστεύει ότι κατά κάποιον τρόπο είναι ακόμα μέλος του ΝΑΤΟ. Τι ακριβώς συμβαίνει με τη συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στη Γεωργία και την Κοντολίζα ε, μια συμφωνία που υπογράφηκε πρόσφατα από ό,τι ξέρετε. εξακολουθεί να επικρατεί η άποψη ότι η Γεωργία μπορεί σύντομα να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτή η άποψη. Ευχαριστώ κύριε Νταφ. Νομίζω ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις ε, είναι ε, ερωτήσεις ε, που μπαίνουν σε βάθος και θα έλεγα λοιπόν για να μπορεί ο κύριος ε, Μορέλ να ε, προλάβει την πτήση του προς τη Νέα Υόρκη να λάβει πρώτα εκείνος ε, το λόγο και μετά θα ακολουθήσει ο κύριος Σάναμπη. Κύριε Μορέλ έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας και την κατανόηση των μελών της Επιτροπής για τα χρονικά πλαίσια που είμαι υποχρεωμένος να τηρήσω. Προετοιμάστε συζήτηση για την εντολή της ε, ΑΜΕΝΙΓ πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Γενικού Γραμματέα σε σχέση με την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά, γιατί οι εμπειρίες μας έχουν μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό και εμείς είμαστε αλληλέγγυοι για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων της Γενέβης. Στην κυρία Ισλέρ Μπεγγέν, Εγώ δεν ε, εξέτασα τα προηγούμενα και τους λόγους για τους οποίους καταλήξαμε σε ένα πόλεμο. Νομίζω ότι ο Πίτερ Σένεμπι με μεγάλη ειλικρίνεια έθεσε το θέμα της ανάγκης αυτοκριτικής για όλους τους φίλους της Γεωργίας. Εγώ βέβαια περισσότερο <clears throat> έχω εστιάσει στο τι έγινε μετά την κρίση αυτή, μετά τον πόλεμο. Για το θέμα τώρα του καθεστώτος το οποίο υπάρχει επιτοπίως. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπα προηγουμένως, έχει καθοριστεί από το Συμβούλιο Υπουργών της 1ης Σεπτεμβρίου. Εμείς καταδικάζουμε την αναγνώριση από τη Ρωσία των υποαπόσχηση περιοχών. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση μετά από τον πόλεμο που είναι πρωτοφανής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η θέση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταδικάζει τη ρωσική αναγνώριση είναι το υπόβαθρο της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, τα μορφώματα αυτά, τα de facto μορφώματα όπως λένε πολλές φορές, ποιο είναι το καθεστώς τους στην πραγματικότητα, η κατάστασή τους. Εμείς θεωρούμε ότι η εδαφική ακαιρεότητα είναι απαραίτητη και βασικό στοιχείο όλων των κρατών στην Ευρώπη. Και εμείς ακολουθούμε αυτήν την γραμμή της μη αναγνώρισης, λέμε ότι έχουμε επαφές με ορισμένες οντότητες χωρίς να τις αναγνωρίσουμε. Μπορείτε να πείτε ότι αυτό είναι νομικίστικο. Όχι, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της διεθνούς πολιτικής. Κάνουμε όσο μπορούμε. Πολιτική εργασία με πολύπλοκες διαδικασίες, για να σας ένα παράδειγμα στη Γενέβη, καταφέραμε όλοι να συνεργαζόμαστε για τα θέματα αυτά και εκτός από την Νικαράγουα δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο, σας το υπενθυμίζω, που να έχει αναγνωρίσει την Απχαζία και την Νότια Οσετία. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι είναι πολυεδρική η πραγματικότητα. Μπορεί να υπάρχει η μία αναγνώριση ακόμα και από χώρε που είναι κοντά στη Ρωσία. Αυτό είναι ένα πολιτικό γεγονός. Επομένως, η πολύπλοκη αυτή κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά τι βλέπει τώρα η Γεωργία για το μέλλον της και την εδαφική της ακαιρεότητα. Εγώ σας παραθέτω αυτά που είπε ο πρόεδρος Σακασφίλη στην έναρξη της ε, Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο μίλησε για το στόχο μιας ειρηνικής επανένωσης της Γεωργίας. Άλλοι στη Γεωργία δεν το βλέπουν έτσι και εδώ πρέπει να είμαστε σαφείς. Και εδώ ο καθένα μπορεί να εκτιμήσει την κατάσταση του εσωτερικού τη Γεωργία όπω θέλει. Υπάρχουν πολλέ εντάσει, αλλά σα είπα τι είπε ο επικεφαλή του Γεωργιανού κράτου. Υπήρξαν και άλλε περιπτώσει οι οποίε ήταν ειρηνικέ και σίγουρα στην περίπτωση τη Γεωργία πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολυπλοκότητα και να συνεχίσουμε τι προσπάθειέ μα ειρήνευση και όχι πολεμικών ενεργειών. Και εδώ έρχομαι και στο ερώτημα του κ. Κασουλίδη. Ναι, δεν είναι μια παγωμένη σύραξη, αλλά όταν πράγματι παγώνει διαπραγματεύσει διαπραγματεύσεις ακολουθεί μια σύραξη. Γι' αυτό χρειάζονται διαπραγματεύσει ενέργεια. Χρειάζεται η εργασία όλων αυτών που βρίσκονται επί για να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όσων των δυνατών πιο φυσιολογική και ομαλή. Σε ό,τι αφορά και τι σχέσει των τοπικών αρχών, είτε είναι αναγνωρισμένε και μη αναγνωρισμένε, προ το καλό των πληθυσμών οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο. Γιατί τον Γενάρη κάνει μείον 10 στου ορεινού όγκου τη Γεωργία και το να ζει σε σκηνές είναι κάτι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο και θέτει σε δοκιμασία τις κοινότητες που έχουν πληγεί από την σύραξη του περασμένου έτους. Επομένως, το θέμα είναι το πρακτέον και αυτό είναι το σύνολο των ερωτήσεων που έχουμε για το μέλλον. Η λογική της Γενέβης είναι να ξεκινήσουμε από την συγκεκριμένη και κατεπίγουσα κατάσταση επιτοπίως. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σταδιακά και αυτά τα οποία πράττουμε είναι το πρώτο στάδιο, να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πιο κατεπίγουσες καταστάσεις και να ομαλοποιήσουμε την πραγματικότητα. Στη συνέχεια θα πρέπει να εδραιώσουμε τις καταστάσεις και από τη στιγμή που έχουμε τις απαραίτητες δομές και υπάρχει μια διαδικασία που αποτελεί ένα μηχανισμό, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πιο μακρόπνο έργο που έχει να κάνει με το πολιτικό καθεστώς και τον διάλογο των συνομιλητών σε σχέση με το μέλλον, με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό θα υπάρξει κάποια λύση. Είναι μια γνωστή λοιπόν αλληλουχία προσπαθειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσανατολίζεται σε μια άμεση λύση, αλλά θέλει να ξεπεράσει τα πρώτα στάδια με την χρησιμοποίηση των πολιτικών δυνατοτήτων μας, η αναζωογόνηση των προσπαθειών μας η κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων και η συνεκτική στάση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι στο άμεσο, στο άμεσο παρόν έχουμε δείξει ότι είμαστε σε θέση να τα κάνουμε όλα αυτά. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, έχουμε πάρα πολλά προσκόμματα τα οποία αναδύονται. Σε κάθε συνεδρίαση στην ε, Γενέβη βρισκόμαστε πάντα στο χείλος της ρήξης ή της αποχώρησης, αλλά όλοι κατανοούν ότι είναι σημαντικές αυτές οι διαπραγματεύσεις. Η συνολική λοιπόν πορεία μας είναι σαφή σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις που πιθανόν να έχει, όπως αναφέρθηκα ε, από τα ερωτήματα από τον κύριο Ζήσκεβιτς. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Το καθεστώς των περιοχών αυτών πρέπει να αντιμετωπιστεί από την διασκέψη της Γενέβης. Τα θέματα των ε, σχέσεων επίσης, αλλά το θέμα και το θέμα των παρατηρητών και της πρόσβασής τους πρέπει να αντιμετωπιστεί στη Γενέβη η, παρουσία, η εκπρόσωψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΑΣΕ και του ΟΗΕ έχει περάσει τα, τη διοικητική γραμμή, έχει πάει στο Σουχούμι, έχει πάει στο Τσίμπαλι. Και εμείς δεν έχουμε αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις όπως ορισμένοι θέλησαν να το κάνουν. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια πολιτική ανταλλαγή απόψεων. Πώς θα φτάσουμε στη μόνιμη και σταθερή ειρήνη μόνο σταδιακά αυτό πρέπει να γίνει με τις επιλογές που θα κάνει η Γεωργία, με τις επιλογές της Ρωσίας και με τις οντότητες αυτές να κατανοήσουν ότι δεν έχουν καμία παγκόσμια αναγνώριση, ότι έχουν μια στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στο ελφός τους και ότι υπάρχει μια άμεση ανάγκη για τους πληθυσμούς τους να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά τους προβλήματα. Ο ΙΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΑΣΕ θα τους διευκολύνουν για την παροχή φυσικού αερίου, την υδροδότηση, την επιστροφή των προσφύγων. Όλα αυτά είναι στην μέση διάθεση. Για το ΝΑΤΟ τελικό ερώτημα, αυτό δεν αφορά την κρίση, Νομίζω ότι αυτό είναι το μακροπρόθεσμο και είναι η ευκαιρία να δώσω το ρολό στον κύριο Σενεμπή και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη της Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την προσοχή σα. Σας ευχαριστώ πάλι κύριε Πρέσβη για την παρουσία σας και για την παρουσίαση της ε, εικόνας που έχετε για τη Γεωργία και ξέρουμε ότι πρέπει να φύγετε και σας ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτηση για τη Γεωργία και τον Νότιο Κάφκασο. Ο κύριος Σάνεμπι ε, συμφωνεί να σχολιάσει περαιτέρω ε, για τις ερωτήσεις που ήδη τέθησαν. Πριν όμως δώσω το λόγο, θα δώσω το λόγο να τεθούν ε, άλλες δύο ερωτήσεις και μετά θα απαντήσει ο κύριος Σάνεμπι. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να είμαι σύντομος, θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Είναι βέβαια αυτονόητο και εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γαλλική Προεδρία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Κατορθώσαμε τουλάχιστον ε, αυτή τη διαδικασία να την διαχειριστούμε κατά κάποιον τρόπο. Υπήρξε λοιπόν μια συμφωνία έξι σημείων. Υπήρξαν ε, προϋποθέσεις ε, Μία από αυτές ήταν η απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων και η επαναφορά του καθεστώτος πριν από την έναρξη των συγκρούσεων. Παρ' όλα αυτά όμως η Ρωσία αναγνώρισε αυτές τις δύο εδαφικές οντότητες και τώρα να δούμε λιγάκι ποιο ακριβώς θα πρέπει να είναι το καθεστώς που πρέπει να επικρατεί. Ο κύριος Μορέλ μας είπε ότι η Ρωσία κάνει βήματα προς την κατεύθυνση επίτευξης στόχου. Αλλά ποιος είναι τελικά ο στόχος, ποιο είναι το καθεστώς ε, που θα έχουν αυτά τα δύο ε, κράτη ή κρατικές οντότητες. Και κατά δεύτερον, τι ακριβώς συμβαίνει με την ε, ειρνευτική αποστολή. Στη Νότια Οσετία είχαμε 1.500 άτομα που εργάστηκαν στην ειρηνευτική αποστολή. Γνωρίζουμε όμως ότι οι Ρώσοι αύξησαν κατά πολύ τον ε, αριθμό των δικών τους ε, των ε, συνεργατών το 1995 υπήρξε μια συμφωνία για αυτή την ειρηνευτική αποστολή και ρωτώ κατά πόσον η συμφωνία αυτή εξακολουθεί να υπάρχει ή μήπως το ρόλο αυτό τον αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μήπως τελικά πρόκειται για δύο διαφορετικές ειρηνευτικές αποστολές. Ο κύριος Ονεσκέβιτς. Έχω τρεις ε, ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά ε, στο καθεστώς της Κασπίας και σε ποιον βαθμό το θέμα αυτό ε, αναχαιτεί στις προσπάθειες ε, κατασκευής ε, αγωγού που θα περνάει από το Τουρκμενιστάν, το Καζακστάν και το Αζερβαϊτζάν. Κατόπιν, ο ρόλος της Γκουαμ, η Γκουαμ παίζει κάποιο ρόλο ή θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο και τέλος, η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν είναι πρόθυμες οι χώρες αυτές να χωρίσουν κάποια εδάφη τους ε, για να είναι πιο ασφαλής η πρόσβαση στον Αχίτσεβα και στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Αυτές είναι οι ερωτήσεις και δίνω τον λόγο στον κύριο Σένεμπι. Πολύ σύντομα σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να θέσω αυτό το ερώτημα για τη Γεωργία. Κύριε Σεμνεύη, <clears throat> μήπως μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο σε σχέση με την κατάσταση του ρωσικού στρατού στην Αυχαζία και την Νότια Οσετία και συγκεκριμένα σε σχέση με τις βάσεις που θέλουν να εγκαταστήσουν εκεί Φαντάζομαι ότι θα είναι βάσεις από τις οποίες δεν θα φύγουν ποτέ. Έχουμε δύο εκθέσεις από τις ε, αντιπροσωπείες, από τις αποστολές που πήγαν εκεί. Ξέρετε αν κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών μπορέσαν να πάνε στην Νότια Σετία και την Απχαζία για να δουν επιτοπίω στην κατάσταση. Και επίσης, συνολικά για τον Νότιο Κάφκασο, πιστεύω ότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Μήπως πιστεύετε ότι παρά την πολιτική γειτονία που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και μια υποχώρηση σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας έκφρασης. Είπατε τι έγινε στο Αζερμπαϊτζάν, ότι παρατάθηκε η εντολή του Προέδρου, ότι αρνήθηκαν τις άδειες σε ραδιοτηλεοπτικές εταιρείε και τα λοιπά στην Αρμενία έχετε πολιτικούς κρατουμένους Έχετε ορισμένους οι οποίοι φαίνεται ότι είναι κρατούμενοι από τις μυστικές υπηρεσίες. Έχετε λοιπόν μια σαφέστερη εικόνα του τι συμβαίνει σήμερα σε αυτές τις χώρες. Επίσης έχουμε την εντύπωση ότι στον Αγκόνο Καραμπάχ υπήρχε μια δυνατότητα να αντιμετωπιστεί και να επιληθεί αυτή η σύγκρουση. Είπατε ότι ίσως θα γίνει κάτι το καλοκαίρι. Μήπως πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ψήγμα ελπίδας να απελευθερωθεί αυτή η περιοχή του Αζερμπαϊτζάν και τι συμβαίνει με την ε, πίεση που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανοίξουν τα σύνορα μεταξύ Αρμενίας και Τουρκίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ο κύριο Σένεμπι τώρα θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μου είπαν ότι έχω 12 λεπτά για να απαντήσω 13, όχι 12, 13. 13 λεπτά έχετε. Θα προσπαθήσω λοιπόν όσο καλύτερα μπορώ να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις και του πρώτου κύρου και του δεύτερου. Όσον αφορά το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρθηκε και έγινε δεκτή ως ε, διαμεσολαβητής και αυτό ε, σε μεγάλο βαθμό λόγω της πολύ καλής εργασίας της Προεδρίας αλλά γενικότερα και λόγω της εικόνας που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια ήπια δύναμη ε, που δίνει μεγαλύτερο βάρος ε, στην πυθό και λιγότερο στην, ε, στον πιθαναγκασμό. Έτσι λοιπόν ήταν θέμα αξιοπιστίας που είχε προκαλέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και αυτό μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βεβαίως παραμείναμε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένε Πολιτείες καθ' όλη τη διάρκεια ε, καταβολής αυτών των προσπαθειών και οι Ηνωμένε Πολιτείε αποτελούν και αυτές ε, μέλος συμμετέχουν στη διαδικασία της Γενέβης. Επίσης και τα Ηνωμένα Έθνη συμμετέχουν ε, στη συζήτηση για την Απχαζία υπάρχει μια σχετική εντολή των Ηνωμένων Εθνών. Και οποιαδήποτε λύση εξευρεθεί θα πρέπει να ε, υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών ε, σχετικά με τον τελικό στόχο. Όσον αφορά τώρα το χάρτη Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Γεωργίας, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο κατά κύριο λόγο έχει ως στόχο να ανταποκριθεί σε πάρα πολλές ανησυχίες ε, σχετικά με την ασφάλεια της ε, γεωργίας που προέκυψαν μετά τον πόλεμο και πολλές ε, προϋποθέσεις που δεν καλύπτονται από τη γεωργία επικράτησε απογοήτευση στη γεωργία γιατί δεν έλαβε ένα πρόγραμμα δράσης. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ακόμα και αν δεν είναι αυτό ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως το πρόσφερε το ΝΑΤΟ, στη τελική ανάλυση είναι κάτι που από κοινού με άλλους παράγοντες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα βοηθήσει στο να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Δεν θα μιλήσω βέβαια εξ ονόματος οποιοδήποτε, αλλά θα ήθελα να πω ότι παραμένει ανοιχτό το θέμα, δηλαδή τι είδους ε, επιπτώσεις ε, υπάρχουν ε, για τις δυνάμεις στη γεωργία. Και, και αυτό είναι κάτι που ετέθη στο χάρτη Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας, αλλά με περιπτώσει δεν είναι ακόμα απόλυτα σαφές για το ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις και των δύο πλευρών και βεβαίως και υποχρεώσεις των ΗΠΑ. Εξάλλου υπήρξαν και κάποια θέματα που αφορούν στη συνεργασία ε, στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν θα προχωρήσω πάρα πολύ στο θέμα αυτό. Κατ' ουσίαν αυτό που έχουμε είναι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία συζητείται στα κράτη-μέλη. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι αυτό είναι ένα τμήμα του πακέτου το οποίο εγκρίθηκε από το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η συμφωνία αυτή διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο γιατί από τη συμφωνία αυτή φάνηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμη να ε, εμπλακεί όχι μόνο στη σύραξη αυτή που είχε ξεσπάσει, αλλά και μακροπρόθεσμα. Έτσι λοιπόν αποδείχθηκε ότι ε, έπρεπε να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των χωρών ε, της Ανατολικής Ευρώπης το γεγονός ότι είχαν ε, και έχουν μια συγκεκριμένη ιστορία έχουν προσδοκίες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή ε, δικές τους περιφερειακές ανησυχίες που δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα. Όσον αφορά τώρα το θέμα των συμφωνιών που έτυχαν διαπραγμάτευσης. Δηλαδή η Συμφωνία περί κατάπαυσης του πυρός και η Συμφωνία της 11 Σεπτεμβρίου κατά πόσον ε, τηρήθηκαν αυτές ε, οι συμφωνίες. Η Συμφωνία της 11 ε, Σεπτεμβρίου αφορά κυρίως στην απόσυρση από τα όμορα κράτη της Γεωργίας και της, της Απχαζίας και της Νότιας Οσετίας. Βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε ρόλο σε αυτή την απόφαση. Ε, το σχέδιο των έξι σημείων ε, έχει σχέση με την ε, κατάπαυση του πυρός αλλά αυτό όπως είπε και ο κύριος Μορέλ είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο των συζητήσεων της Γενέβης. Όσον αφορά τώρα το καθεστώς ε, αυτών των εδαφών, αυτό δεν υπάρχει προς το παρόν στην ε, ημερήσια διάταξη. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιοδήποτε άλλος ε, παράγων στηρίζει την αναγνώριση από πλευράς Ρωσίας της ανεξαρτησίας της Απχαζίας και της Νότιας Οσετίας. Απλά βρισκόμαστε τώρα σε μια φάση όπου είναι πολύ νωρίς να εισάγει κανείς το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Αν γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι οι σημαντικές συζητήσεις που γίνονται τώρα για θέματα των προσφύγων, της ασφάλειας, της ε, αποφυγής ατυχημάτων. Οι ε, συζητήσεις αυτές θα καταστούν πολύ πιο δύσκολες, αν θέλετε, έως και αδύνατες. Τώρα, ας δούμε τι ρόλο θα διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στη σύγκρουση αυτή, κυρίως στη Νότια Οσετία, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα ε, διδραματίσει ειρηνευτικό ρόλο, θα συμμετάσχει στην ειρηνευτική αποστολή που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές. Δεν είναι εύκολο να δώσει κανείς απάντηση στο ερώτημα αυτό, προς το παρόν τουλάχιστον. Δεν ε, προβλέπονται άμεσα σχέδια για την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να αναλάβει αυτό τον ειρηνευτικό ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να αναθεωρήσει ε, τη δουλειά ε, της ειρνευτικής αποστολής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Σεπτέμβρη αυτού του έτους όταν θα εκπνεύσει αυτή η αποστολή θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία να δούμε πώς μπορεί, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να είναι παρούσα επιτόπου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ληφθούν βέβαια υπόψη και οι συζητήσεις που θα λάβουν χώρα στη Γενέβη. Όσον αφορά τώρα του ε, τους στόχους της Ρωσίας σε όλη αυτή τη σύγκρουση, νομίζω ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα. Υπάρχουν ε, διάφορα επίπεδα της σύγκρουσης και αυτό είναι επίσης κάτι που πρέπει να έχουμε κατά νου όταν θα σχεδιάσουμε την απάντησή μας ε, στην σύγκρουση αυτή. Έχουμε πρώτα απ' όλα την ε, διακοινωτική σύγκρουση ανάμεσα ε, στην Απχαζία και τη Γεωργία και αυτή η διένεξη είναι κατ' ουσίαν και η ρίζα του προβλήματος. Είναι μια διένεξη η οποία ε, κατά κάποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για την αντιπαράθεση ανάμεσα στη Γεωργία και τη Ρωσία. Υπάρχουν κάποια στοιχεία ε, εδαφικών, ε, εδαφικής ε, αμφισβήτησης, ακόμα και προσωπικών σχέσεων των δύο ηγετών. Υπάρχουν στοιχεία που έχουν σχέση με στρατηγικό ανταγωνισμό και αυτά ξεπερνούν το στενό πλαίσιο του Νότιου Καυκάσου. Όσον αφορά τώρα στο καθεστώς της ε, Κασπίας, κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσον ε, θα μπορέσουν, θα καταστεί δυνατόν να συμφωνήσει κανείς σε, σε θέματα Κασπίας. Κοιτάξτε, ε, υπάρχουν κάποια εμπόδια όσον αφορά τους ε, αγωγούς ε, και κάποια άλλα στοιχεία υποδομής ε. Πάντως αυτό που παίζει ρόλο είναι οι συζητήσεις Αζέρων και Τουρκμένων ε, σχετικά με τον αγωγό κατά πόσον ε, ε, θα μπορούσε αυτός ο αγωγός να συνδυαστεί και με τον αγωγό που διασχίζει το Αζερμπαϊτζάν. Μιλάμε για ένα αναγωγό βέβαια που θα είναι 60-70 χιλιόμετρα. Δεν θα χρειάζεται να ε, διασχίζει ολόκληρη την Κασπία ε, καθότι τα κοιτάσματα του Τουρκμενιστάν είναι κοντά σε αυτά του Αζερμπαϊτζάν. Πάντως ε, θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια να συνδεθούν αυτοί οι δύο αγωγοί και εγώ ε, πιστεύω ότι είναι προς όφελος του Τουρκμενιστάν ε, το να θελήσει να ε, διαφοροποιήσει τις δυνατότητες που έχει. Η πλευρά των Αζέρων πάντως ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα όσον αφορά το ρόλο της Γκουαμ Πρόκειται για μια οργάνωση η οποία βέβαια είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, μεταπτώσεις. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια οργάνωση Μάλλον το παλιό λέει ο μιλητή. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Δεν συμμετέχουν στην ΚΟΑΜ όλες οι χώρες της περιοχής. Και η ΚΟΑΜ ε, έχει κατηγορηθεί ότι είναι περιοριστική. Με την έννοια ότι ενδιαφέρεται ε, περισσότερο ε, για ε, μια αντίσταση κατά της Ρωσίας. και αναπτύσσεται βέβαια με την έννοια ότι έχει συστήσει ε, μια γραμματεία στο Κίεβο. Ε, θα ε, ασχοληθεί με πάρα πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών θεμάτων. Και θα μπορούσε πράγματι η Γκουαμ να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, να παίξει ρόλο και έτσι ώστε να μπορέσει η Γκουαμ να προβάλλει ε, κάποια σημεία της ε, ημερήσιας ε, διάταξης που θα ξεπερνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη στενή έννοια και θα αφορούν περισσότερο τους εταίρους μας προς Ανατολάς. Όσον αφορά το Αγκόρνο Καραμπάχ, ε, τέτοιο ερώτημα κατά πόσον είναι πρόθυμες ε, οι Αρμενοί και το Ζερμπετζάν να ανταλλάξουν εδάφη. Κοιτάξτε, αυτό δεν συζητήθηκε τώρα, ε, συζητήθηκε κατά παρελθόν και όταν συζητήθηκε αποδείχθηκε ένα ιδιαίτερα επίμαχο θέμα. Είμαστε λοιπόν πολύ μακριά από το να συμβεί κάτι τέτοιο. Και Αυτό τη στιγμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι μια διαφορετική έννοια Δηλαδή θέλουμε να αποσυρθούμε από όλα τα κατεχόμενα, να υπάρξει απόσυρση στρατευμάτων από όλα τα κατεχόμενα εδάφη, να υπάρχει μια, ένα ενδιάμεσο καθεστώς για τους ε, πρόσφυγες του Ναγκόρνο Καραμπάχ και να ε, πάυσει πλέον να επικρατεί αυτή η ασάφεια τουλάχιστον για το μέλλον. Αυτή τη λύση αναζητάμε τώρα. Όσον αφορά τώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ε, Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Εδώ θα μπορούσε κανείς να πει πάρα πολλά και με πολλές λεπτομέρειες αλλά φοβάμαι ότι δεν έχουμε πια χρόνο για να μπούμε σε λεπτομέρειες. Εγώ πάντως θα ήθελα να πω ότι το θέμα των ατόμων που βρίσκονται υπό περισμό, δηλαδή η αντιπολίτευση στην ε, Αρμενία και οι δημοσιογράφοι στο Αζερβαϊτζάν, αυτό το θέμα θα μπορούσε πολύ εύκολα να λυθεί μέσα από αποφάσεις από τους ε, αρχηγούς ε, κρατών. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό ε, το όλο θέμα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Όσο υπάρχουν τα άτομα αυτά, θα δημιουργούν πρόβλημα στις σχέσεις μας. Και νομίζω ότι τούτο το γνωρίζουν οι ηγεσίες και των δύο κρατών. Για την πρόσβαση προς την Απχαζία και την Νότια Οσετία σε ό,τι αφορά τις διεθνείς αποστολές ερευνητικού χαρακτήρα. Είναι πρόβλημα αυτό. Όχι μονάχα ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν πρόσβαση στην Απχαζία και την Νότια Οσετία. Ακόμα και οι διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και κατά πάσαν πιθανότητα οι διάφορες ομάδες που προσπαθούν να κάνουν έρευνες είτε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από την πλευρά των ΜΚΟ έχουν προβλήματα. Ανησυχητικό είναι αυτό, διότι η κατάσταση είναι μία κατάσταση όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα του υπόλοιπου πληθυσμού των Γεωργιανών στις ε, υποαπόσχησης περιοχές είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί τα μάλα. Στην περιοχή του Γκάλι στην Απχαζία και το Αχαγκόλι στην Νότια Οσετία υφίσταται μεγάλες πιέσεις ο γεωργιανός πληθυσμός εκεί. Τα σύνορα γίνονται όλο και πιο στεγανά. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα για τον τοπικό πληθυσμό, ο οποίος στο παρελθόν διακινεί το ελεύθερα. Ε, στην περιοχή αυτή υπάρχουν περιοχές επιβολής μιας ρωσικής έκδοσης ρωσικών διαβατήριων, όλα αυτά συγκροτούν ένα περιβάλλον το οποίο φαίνεται να είναι εκφοβιστικό για τον τοπικό πληθυσμό. Μια σημαντική στρατιωτική παρουσία των Ρώσων επίσης στην περιοχή και αυτό είναι το πιο καλόβουλο αν θέλετε τμήμα της παρουσίας αλλά ιδίως στην περιοχή του Αχαγούν υπάρχει και σημαντική παρουσία πολιτοφυλακών της Νότιας Οσετίας η οποία είναι πολύ προβληματική σε σχέση με την συμπεριφορά της και είναι εκτός ελέγχου. Νομίζω ότι απήντησα σε όλα αυτά τα ερωτήματα και μου είπαν ότι έχουν περάσει στα 13 μου λεπτά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλα αυτά που είπατε. Ήσασταν πάρα πολύ στην παρουσίαση των πολυπλοκοτήτων της κατάστασης και δυστυχώς δεν είναι η τελευταία φορά που πρέπει να συναντηθούμε για να εξετάσουμε αυτή την κατάσταση. Βασιζόμαστε λοιπόν στην συνέχιση αυτού του διαλόγου μαζί σας με την εμπειρογνωμοσύνη που έχετε για τα γεγονότα στο Νότιο Κάφκασο, τη Γεωργία κτλ. Όχι μόνο για τα θέματα που προκύπτουν μετά από τον πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά και για τα στρατηγικά θέματα που μας ενδιαφέρουν σε αυτή την τόσο δύσκολη και κομβική περιοχή της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ λοιπόν, λοιπόν πάρα πολύ και ελπίζω να σας ξαναδούμε σύντομα. Και τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο θέμα και θα ήθελα να ε, δώσω την προηγούμενη στον κύριο Ρότσεκ.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 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με το δεύτερο σημαντικό θέμα στην σημερινή ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Φουαρέ, ο οποίο είναι ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και επικεφαλή της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της ε, Μακεδονίας. Σα καλωσορίζουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι την τελευταία φορά που ήσασταν εδώ ήταν το 2008, πριν από ένα χρόνο. Έκτοτε είχαμε εκλογέ στα Σκόπια, είχαμε έχουμε ένα νέο πρόγραμμα, μια νέα έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στο οποίο πρόγραμμα αναφέρονται κάποιες ε, θετικές εξελίξεις, ε, παραμένουν όμως ακόμα αρκετές προκλήσεις και υπολείπεται ακόμα πολλή δουλειά. Έχοντας λοιπόν κατά νου αυτές τις εξελίξεις. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρέσβη κύριο Φουαρέ, ο οποίος ε, έχει 15 περίπου λεπτά για να κάνει την αρχική εισήγηση και βεβαίως ε, κατόπιν θα ακολουθήσουν ερωταπαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής για το ότι είχαν την ε, καλοσύνη να με προσκαλέσουν σε αυτή τη συνάντηση. Έχει γίνει πλέον πεπατημένη παράδοση από τότε που ανέλαβα το αξίωμά μου ε, να ε, εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Μακεδονία πριν από τρία χρόνια. Έχει γίνει παράδοση να έρχομαι σε αυτή την Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και τον κύριο Έρικ Μάια και τους ε, υπόλοιπους συναδέλφους για το ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στη χώρα και προετοίμασαν μάλιστα και το ψήφισμα αυτό το οποίο πρόκειται να συζητηθεί και να ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2008 ήταν αναμφίβολο αμφίβολα μια δύσκολη χρονιά για την πρώην δημοκρατία της, ε, τη Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ε, είδαμε ότι υπήρξαν κάποιες προϋποθέσεις ε, οι οποίες ανεφέρθη ότι εάν πληρούνται από τη χώρα τότε θα μπορέσει και η Επιτροπή να κάνει μια σύσταση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Όπως γνωρίζετε, οι εκλογές το 2008 ε, ήταν ε, κόλαφος για τη χώρα, γιατί χαρακτηρίστηκαν από ε, ταραχές και ανομαλίες κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Το συμπέρασμα που εξήχθη είναι ότι οι εκλογές αυτές δεν καλύπτουν τις διεθνείς προδιαγραφές. Κατόπιν ακολούθησε τον Ιούλιο του 2008 ε, μια έκτακτη διαδικασία έτσι ώστε να ε, περάσει νομοθετικές πράξεις και δυστυχώς αυτή τη φορά ε, τα νομοσχέδια αυτά απεκλείστησαν και μποϊκοταρίστηκαν από την αντιπολίτευση. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι παρόλα αυτά έλαβαν χώρα σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσει αυτές περιλαμβάνονται στην έκθεση προόδου την οποία παρουσίασε την 5η Νοεμβρίου Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση αυτή ορίζει τους τομείς στους οποίους εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και τομείς τους οποίους θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω θα έλεγα ισχυρές παρεμβάσεις από πλευράς της κυβέρνησης. Η εκθεση αυτη οριζει τους τομεις στους οποιους εξακολουθουν να υπαρχουν σοβαρα προβληματα και τομεις στους οποιους θα πρεπει να υπαρξουν περαιτερω θα ελεγα ισχυρες παρεμβασεις απο πλευρά της κυβερνησης η κυβερνηση δεχεται την έκθεση πρόοδου σαν μια αξιολόγηση της γενικότερης προόδου και αυτό είναι κάτι το ενθαρρυντικό. Δέχονται δηλαδή αυτά που λέμε. Επίσης η κυβέρνηση υιοθέτησε το λεγόμενο Blueprint for National Action το οποίο ε, περιλαμβάνει τους βασικούς άξονες τους οποίους η κυβέρνηση στα Σκόπια θα προωθήσει και θα προωθήσει επίσης και μια σωστή καταγραφή του ρυθμού εφαρμογής της νομοθεσίας η οποία έχει ήδη υιοθετηθεί. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε και από τον Αντιπρόεδρο Μποτσεύσκη στις 2 Ιανουαρίου σε μια συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής στα Σκόπια. Επανέλαβε ο κύριος Μποσένσκι τις τρεις προτεραιότητες για το 2009. Πρώτον, υποστήριξη των ευρωπαϊκών στόχων μέσω της πλήρους εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου για την εφαρμογή των συστάσεων της εκθέσεως προόδου και δεύτερον εκπλήρωση των βασικών πολιτικών κριτηρίων ιδιαίτερα σε σχέση με τις επερχόμενες τοπικές και βουλευτικές εκλογές και προεδρικές συγγνώμη εκλογές όπως επίσης και προώθηση του διαλόγου ανάμεσα στους πολιτικούς θεσμούς. Επίσης συνέχιση των προσπαθειών για την απελευθέρωση του καθεστώτος χορήγησης θεωρήσεων, όπως επίσης και για την διαπίστευση των υπηρεσιών για την χρήση των πιστώσεων από πλευράς του προενταξιακού μέσου. Πρόκειται για μια συνολικά θετική παρουσίαση από πλευράς της κυβέρνησης, είναι κάτι το οποίο καλωσορίζουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεχίζεται η προσπάθεια από, μια κυβερνητική συνασπιστη... από ένα σχήμα συνασπισμού το οποίο προς το παρόν προχωρά με επιτυχία και ελπίζω να συνεχιστεί η επιτυχία αυτή και μετά από τις προεδρικές εκλογές. Ποιες είναι τώρα οι βασικές προκλήσεις που έχει μπροστά της η Καταρχάς οι εκλογές. Οι εκλογές είναι η πιο σημαντική πρόκληση. Έχουν μείνει δύο μήνες πριν από τις τοπικές δημοτικές δηλαδή εκλογές και τέσσερις μήνες ε, και τρεις μήνες μάλλον για τις προεδρικές οι οποίες θα γίνουν στις 22 Μαρτίου και 5 Απριλίου θα γίνει ο δεύτερος γύρος για τις προεδρικές. Θα πρέπει να υπάρξει μια τεράστια προσπάθεια από τις δικαστικές αρχές να ολοκληρωθούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες εναντίον αυτών οι οποίοι διέπραξαν ανομίες στις εκλογές του 2008. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση έτσι ώστε να καταργηθεί αυτό το κλίμα ατιμορρησίας το οποίο ίσχυε μέχρι το 2008. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρης εφαρμογή όλων των συστάσεων τις οποίες έχει κάνει η ομάδα παρατηρητών του ΟΑΣΕ Υπάρχει επίσης και η εκλογική επιτροπή η οποία έχει νέα σύνθεση και θα έχει την πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να διασφαλίσει ότι τα πάντα θα προχωρήσουν ανεμπόδιστα στα πλαίσια μιας περίπλοκης εκλογικής διαδικασίας λαμβάνοντας υπόψη ότι θα γίνουν ταυτόχρονα δύο εκλογές. Παράλληλα, η σύνθεση της τοπικής εκλογικής επιτροπής των τοπικών εκλογικών επιτροπών, 2.000 σε όλη τη χώρα, στο παρελθόν απαιτελούνται από πέντε υπαλλήλου. Τώρα όμως θα αποτελούνται από τρει υπαλλήλου και από δύο εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Αυτό απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση για τα μέλη των επιτροπών αυτών, γιατί αυτές οι επιτροπές θα επιβλέψουν την λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας την ημέρα των εκλογών θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι δηλαδή ότι όλοι οι κανόνες θα γίνουν πλήρως σεβαστοί και αυτό θα πρέπει να γίνει μακράν κάθε πολιτικής επεμβάσεως. Ταυτόχρονα έχει μεγάλη σημασία το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο θα να έχει τους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς πόρους, έτσι ώστε να παρακολουθεί τη χρήση των μέσων ενημέρωσης και να διασφαλίσει την μη κατάχρηση των μέσων ενημέρωσης από ένα από τα πολιτικά κόμματα. Και τα θέματα ασφαλείας επίσης δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν. Στοχεύουμε σε ένα πρόγραμμα ασφαλείας το οποίο έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση και θα το καταθέσει σύντομα. Στα πλαίσια επίσης της συνεργασίας μας σε επίπεδο υποστήριξης των αστυνομικών δυνάμεων και μεταρρύθμισης των αστυνομικών δυνάμεων παρέχουμε εκπαίδευση για την αστυνομία της χώρας για τις εκλογικές διαδικασίες ειδικά Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ώστε οι εκλογές αυτές να σεβαστούν όλα τα διεθνή επίπεδα και αυτό θα εξαρτηθεί από την ίδια τη συμπεριφορά των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ηγετών και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και κατά τη διάρκεια της ημέρας των εκλογών. Και αυτό θα καθορίσει αν στο τέλος της διαδικασίας θα κρυθούν από πλευράς μας οι εκλογές αυτές δίκαιες και δημοκρατικές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το συγκρουσιακό πνεύμα το οποίο χαρακτήριζε τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς ηγέτες πριν από τις εκλογές του 2008 συνεισέφερε τα μάλα στις ανομίες οι οποίες διαπράχθησαν εκείνη την περίοδο. Και αυτό οδηγεί σε μία άλλη σημαντική σύσταση από πλευρά της εκθέσεω της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ανάγκη δηλαδή για έναν ισχυρό πολιτικό διάλογο χωρίς εξαιρέσει, χωρίς αποκλεισμού σε πνεύμα συνεργασίας, σε πνεύμα συνένεσης, κάτι το οποίο έλειπε τα προηγούμενα χρόνια από τη χώρα υπήρξε μια συνάντηση ηγετών όλων των πολιτικών ηγετών που οργανώθηκε από τον Πρωθυπουργό τις τελευταίες εβδομάδες μια πολύ θετική συνάντηση και ελπίζω ότι εφόσον συνεχίσουμε στο πνεύμα αυτής της συνάντησης θα υπάρξει περαιτέρω πολιτικός διάλογος. Συνεχίζουμε επίσης και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας Πλαισίου της Αχρίδας. Είναι θα έλεγα βασικό στοιχείο της προώθησης των συνθηκών συμβίωσης της πολυεθνικής αυτής κοινωνίας. Πρέπει να υπάρξουν λοιπόν περαιτέρω ισχυρές προσπάθειες ιδιαίτερα για την επίτευξη της ισότιμης αντιπροσώπευσης της ε, κοινότητας, των, των κοινοτήτων των μειονοτικών. Πολλά μένει να γίνουν έτσι ώστε η τουρκική κοινότητα, η κοινότητα των Ρωμά να έχουν και αυτές πρόσβαση ε, στην ε, δημόσια διοίκηση να μπορούν να εργάζονται στη δημόσια διοίκηση, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της συμφωνίας πλαισίου της Αχρίδας είναι η εκπαίδευση. Υπάρχει ανησυχία μεγάλη για τις διαχωριστικές γραμμές στην παιδεία που εμφανίστηκαν τους τελευταίους μήνες και που είναι αντίθετες με το πνεύμα της Συμφωνίας Πλαισίου Αχρίδας και εμείς ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση να εφαρμόσει τις συστάσεις ε, και του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως επίσης και του ΟΑΣΕ που θα επισκεφθεί τα Σκόπια σύντομα. Στο δικαστικό έχουν ληφθεί νομοθετικά μέτρα αλλά θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο εφαρμόζονται έτσι ώστε να υπάρξει η πραγματική εμπιστοσύνη της κοινή γνώμης στην δίκαια κρίση της δικαστικής εξουσίας, κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Το σοφρονιστικό σύστημα δεν έχει προσεχθεί ιδιαίτερα από την κυβέρνηση παρά τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και υπάρχουν πολλά τα οποία μένει να γίνουν για να αντιμετωπιστούν κάποιες ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στα σοφρονιστικά καταστήματα Παράλληλα η καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να ενισχυθεί και αυτό θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα κόμματα να μην εμπλέκονται ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε την προεκλογική περίοδο. Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερος γιατί κάθε φορά που υπάρχει νέα κυβέρνηση υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα υπογραμμίσω δύο επιπλέον τομείς οι οποίοι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από πλευρά της κυβέρνησης. Πρώτον, η κοινωνία των πολιτών. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αφιερώσει πολύ περισσότερες προσπάθειες για την εμπλοκή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Είναι τα μάτια και τα αυτιά του κοινού και πραγματικά ο ρόλος τους είναι να κάνουν κριτική και θα πρέπει η κυβέρνηση να ακούει την κριτική αυτή την οποία υφίσταται. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν η κυβέρνηση να προωθήσει μια πιο ανοιχτή πολιτική διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και να μην προσπαθεί να περιθωριοποιήσει τις οργανώσεις των πολιτών οι οποίες ασκούν κριτική αλλά το κάνουν αυτά στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες στη χώρα. Και ο δεύτερος τομέας, ο οποίος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, είναι τα μέσα ενημέρωσης. Σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ξεκάθαρη. Τα μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να υφίστανται πολιτικές παρεμβάσεις ισχυρότατες Πάρα πολλοί σταθμοί τηλεοπτικοί είναι είναι, ανήκουν σε ιδιώτες που συνδέονται με πολιτικά κόμματα όμως και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε και να πείσουμε και την κυβέρνηση ότι έχουν κάθε συμφέρον να διασφαλίσουν ελεύθερα μέσα ενημέρωσης γιατί δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να δοθούν εγγυήσεις για το πνεύμα διαλόγου και συνένεσης και δεν θα πρέπει να στιγματίζουν τα μέσα ενημέρωσης και να τα περιθωριοποιούν αν ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Μέσω ακριβώς αυτής της δεκτικότητας και της αποδοχής της κριτικής η κυβέρνηση προωθεί τον διάλογο, προάγει τον διάλογο, προάγει το πνεύμα συνεργασίας, προάγει το πνεύμα συνένεσης ανάμεσα σε όλους εταίρους της κοινωνίας. Δύο τελευταία σημεία. Πρώτον, σχετικά με τη χορήγηση θεωρήσεων. Εδώ υπάρχει ένας τομέας όπου η χώρα έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες για την εκπλήρωση για να φτάσουν εν πάση περιπτώσει στα επίπεδα τα οποία θα οδηγήσουν με τη σειρά τους την απελευθέρωση από το καθεστώς θεωρήσεων. Πράγματι έχουν γίνει ιδιαίτερες προσπάθειες, θα πρέπει να κρυθούν οι προσπάθειες αυτές και οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να αξιολογηθούν και αν δουν ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις έχουν επιτευχθεί τότε αυτό θα πρέπει να γίνει αντικείμενο αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η χώρα να μπορέσει να πετύχει τον στόχο πλήρους απελευθέρωσης του καθεστώτος θεώρησης. Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα προς την κοινή γνώμη το οποίο θα λέγεται ότι αναγνωρίζουμε τα βήματα προόδου τα οποία έχουν πετύχει. Και ένα τελευταίο σημείο, θα ήθελα να εκφράσω την αξιολόγησή μου για τις προσπάθειες ε, της ε, Επιτροπής της Μικτής Κοινοβουλευτικής υπό την Προεδρία των κυρίων Τρακατέλη και Σπασενόφσκι. Ήρθαν το φθινόπωρο στα Σκόπια και θα ήθελα να υποστηρίξω τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της συνεργασίας και ανάμεσα στις γραμματείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, της ε, Εθνοσυνέλευσης της ΦΥΡΟΜ. Ε, Αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την Εθνοσυνέλευση της χώρας να εκπληρώσει το ρόλο της σαν δημοκρατικό όργανο πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Εγώ και οι συνάδελφοί μου στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προωθήσουμε και να ενθαρρύνουμε τις μεταρρυθμίσεις όταν αναφύονται προβλήματα ερχόμαστε σε επαφή με την κυβέρνηση, τα σημειώνουμε και ελπίζουμε ότι τελικά η χώρα θα περάσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας ένταξης. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αρχική σας παρουσίαση αυτή. Κανονικά θα έδινα το λόγο στον εισηγητή μας τον κύριο Μάιερ, αλλά ο κύριος Γκάλερ πρέπει να φύγει στις 5 να πάει στη συνέλευση των Προέδρων και όλος εξαιρετικός θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλερ για ένα ερώτημα και μια απάντηση και μετά θα πάρει το λόγο εισηγητής ο κύριο Μάιερ. Σας ευχαριστώ πολύ για το θέμα της χορήγηση των θεωρήσεων. Αναφερθήκατε στο τέλος της παρέμβασής σας. Και θέλω να ρωτήσω, ποιοι είναι οι ουσιαστικοί λόγοι γιατί δεν είναι δυνατόν να αρθούν οι προϋποθέσεις ε, για τις θεωρήσεις. Υπάρχει η Συμφωνία Επανένταξης και επανεισδοχής και υπάρχουν επίσκετα χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν ε, δεν μπορώ να φανταστώ άλλους ε, σημαντικούς λόγους εμπόδια Μήπως μπορείτε να μας ε, πείτε τι ακριβώς αναζητούν να βρουν αυτή τη στιγμή οι εμπειρογνώμονές σας και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρωθούν οι έρευνες των εμπειρογνωμόνων. Και εν πάση τελική πότε οι Μακεδόνες θα αποκτήσουν ε, τη δυνατότητα εισδοχής χωρίς θεώρηση. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, ε, υπάρχει μία αποστολή από τα κράτη-μέλη που είναι επιτόπου και όλοι αυτοί εξετάζουν όλες τις πτυχές ε, της μεταρρύθμισης που είναι απαραίτητη για την ε, χορήγηση των θεωρήσεων. Και το θέμα των βιομετρικών διαβατηρίων, η χώρα έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε σχέση με άλλες χώρες περιοχής. Υπάρχει και το θέμα της διαχείρισης, ολοκληρωμένης διαχείρισης των χινόρων, δηλαδή δηλαδή η χώρα να κάνει ικανοποιητικούς ελέγχους στα σύνορα όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Όταν λοιπόν θα τελειώσει αυτή η διαδικασία θα ακολουθήσει το Φεβρουάριο μια δεύτερη αποστολή εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσει και άλλα θέματα. Και στο τέλος ε, θα είναι δυνατόν να αξιολογηθεί κατά πόσο καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις ή όχι. Πάντως η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα τέλη Νοεμβρίου ήταν θετική. Αναγνωρίστηκαν τα ε, επιτεύγματα, τα θετικά σημεία. Εντοπίστηκαν ε, κάποια ε, προβλήματα κυρίως στην ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και αυτό το εξετάζουν τώρα οι εμπειρογνώμονες. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί η διαδικασία τότε η Κομισιόν θα αξιολογήσει τις πληροφορίες που θα έχει συγκεντρώσει και θα καταθέσει την πρότασή της. Εμείς βέβαια εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι κάθε χώρα κρίνεται από αυτά που έχει επιτύχει και εάν τελικά η αξιολόγηση της Κομισιόν επισημαίνει ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν με επιτυχία, τότε θα πρέπει να ε, συσταθεί η ε, χορήγηση καθεστώτος ελεύθερου από θεωρήσεις για την Μακεδονία. Δεν έχω κατά νου κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πάντως η έκθεση της Κομισιόν αναφέρει ότι ελπίζουμε κατά τη διάρκεια του 2009 ε, και εμεί θα είμαστε θέση να ε, εξετάσουμε, να τοποθετηθούμε. Εξαρτάται βέβαια και από το Συμβούλιο, αλλά και εμείς ε, πιστεύουμε, όπως και εσείς, το γοργόν και χάρη να έχει. Ευχαριστούμε πολύ για την απάντησή σας. Ο κύριος Μάγερ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε βρισκόμαστε το 2009. Το 2009 είχε λυθεί η απόφαση να δοθεί το καθεστώς της υποψήφιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι πολλά κόμματα τα οποία πρέπει να γίνουν σε επίπεδο διαπραγματεύσεων, αλλά αυτή η διαδικασία διαπραγματεύσεων ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Κάθε συζήτηση που γίνεται σε ετήσιο επίπεδο για την πρόοδο της χώρας αυτής στον δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά πέντε κύριος κεφάλαια. Καταρχήν, ποιε είναι οι ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν για να γίνει η Πουδουγουμού μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λειτουργία της Δημοκρατίας, εδώ αναφέρθηκε ο κύριος Φουάρε για το θέμα αυτό, και υπάρχουν και ζητήματα τα οποία αναφέρονται στο ψήφισμα μου. Τα θέματα της δικαιοσύνης, το περιβάλλον, δικαίωμα εργασία, υποδομές, ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να βρούνε μια λύση, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να ληφθούν ορισμένες πρόνοιες. Επίσης έχουμε και το γεγονός, το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, συζητήσαμε για τα θέματα αυτά με τις ε, παραγωγικές τάξεις και την, θέλησαμε να έχουμε την άποψή τους για το, τα ζητήματα αυτά. Ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσει κανείς είναι πότε θα αρχίσουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Όπως γίνονται αυτή τη στιγμή με την Κροατία, πιο με πιο βραδύ ρυθμό με την Τουρκία, αλλά για τις χώρες αυτές στην Κροατία και την Τουρκία έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Είναι διαπραγματεύσεις οι οποίες μπορεί να χρειαστούν 6 με 8 χρόνια μετά από την έναρξή τους, ώσπου να φτάσουν στην τελική ένταξη. Πέρσι, έλαβαν χώρα τα γεγονότα που γνωρίζουμε όλοι για κατά τη διάρκεια των εκλογών και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα προκύψουν νέες καθυστέρησεις που θα προσθεθούν στις ίδιες υφιστάμενες. Αν γίνουν σωστά και με τον κατάλληλο τρόπο οι εκλογές του Μαρτίου, όπως και οι προηγούμενες ε, εκλογές, νομίζω ότι είναι φανερό ότι η στάση της κυβέρνησης θα είναι να προχωρήσει χωρίς να λάβει υπόψη ενδεχόμενες ατασταλίες θα έχει λάβει χώρα μια μερική εκλογή του Κοινοβουλίου το οποίο έχει μόλις αναλάβει το νέο Κοινοβούλιο της ε, εξουσίας του και εδώ έχει διατυπωθεί η άποψη ότι υπάρχουν ε, υπήρξαν παρεμβολές στο έργο του Κοινοβουλίου. Επίσης, οι σχέσεις με τις γειτονικές χώρες έχουν επίπτωση στις διαπραγματεύσεις και στο, στην έκβαση των διαπραγματεύσεων και αυτά τα προβλήματα οδηγούν σε περαιτέρω καθυστερήσεις. Το κείμενο αναφέρει επίσης ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία θα είναι ικανοποιητική για όλους σε ό,τι αφορά τις ε, διαφορές με άλλα κράτη. Δυστυχώς δεν υπήρξαν πολλές πρόοδοι στον τομέα αυτό. Ο κύριος Νίμιτς, ο οποίος είναι ο διαπραγματευτής ε, και είναι σε επαφή με τη μακεδονική και την ελληνική κυβέρνηση, δεν έχει καταφέρει να βρει κάποια λύση. Οι θέσεις των δύο χωρών είναι αποκλίνουσες, υπάρχει μια στάση διστακτική και παρελκυστική. Δεν έχουμε καταλήξει λοιπόν σε καμία λύση. Αν καταλήξουμε όμως σε μια λύση, δεν θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις. Υπάρχει και το θέμα των προξενικών θεωρήσεων που ανέφερε ο κ. Φουαρέ. Είναι πολύ σημαντικό τι θα πρέπει να γίνει καταρχήν μέσα στην ίδια τη χώρα της Μακεδονίας. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ε, βιομετρικών διαβατηρίων. Είναι πολύ δάπανα βέβαια αυτά τα διαβατήρια αυτή τη στιγμή και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Υπάρχει το θέμα των συνόρων με το κοσυφοπαίδιο και εκεί χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες. Και υπάρχουν επίσης και οι φόβοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε, που έχουν εκφραστεί σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών για το κατά πόσο θα πρέπει να αρθούν ορισμένες ε, μορφές περιορισμών. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να υπάρξει ελεύθερη πρόσβαση για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ίσχυαν οι κανόνες αυτοί με την πρώην Ιουκοσλαβία. Πρέπει όλα αυτά να εφαρμοστούν για να μην υπάρχουν εμπόδια σε ό,τι αφορά την χορήγηση προξενικών θεωρήσεων. Επίσης, η εφαρμογή της Συμφωνίας Σαχρίδας πιστεύω ότι έχουν υπάρξει πρόοδοι, ιδίως σε ό,τι αφορά το αλβανικό στοιχείο που εκπροσωπείται τώρα και στην κυβέρνηση της Πουδογουμού έχουν ε, ληφθεί απαραίτητα μέτρα και πρόνοιες για την ισότητα των δύο βασικών γλωσσών στη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε όμως και ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στις δημόσιες ε, υπηρεσίες και στο δημόσιο μηχανισμό και επίσης η εκπροσώπηση των μικροτέρων μειονοτήτων. Χρειάζονται πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν για να επιτύχουμε την πλήρη ισότητα όλων των συνιστοσών του πληθυσμού. η έκθεση αυτή έχει τύχει περίπου 80 τροπολογιών, 50% περισσότερες από την προηγούμενη φορά. Δεν βλέπω να υπάρχουν τεράστιες διαφορές απόψεων. Πολλές από τις τροπολογίες επικαλύπτονται και κάνουμε προσπάθειες να μειώσουμε αυτή τον αριθμό των τροπολογιών με συμβιβαστικές θέσεις. Σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι υπάρχει συμφωνία των πολιτικών ομάδων και δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να περιμένουμε μεγάλες εκπλήξεις στον τομέα αυτό και υπάρχουν και πολλά στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν σε χωριστές ψηφοφορίες ή ψηφοφορίες κατά μέρη γιατί υπάρχουν και διαφορές αποχρώσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ποια είναι τα θέματα τα οποία ακόμα εκκρεμούν Καταρχήν, η γενική αντιμετώπιση για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα δυτικά Βαλκάνια, αν πρέπει να εκφράσουμε μια άποψη για το θέμα αυτό ή όχι, όπως υποστηρίζω εγώ. Επίσης χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσέγγιση με τη Σερβία, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μειώσει την προσοχή η οποία αποδίδεται στη Μακεδονία γιατί μετά από το 2005 η χώρα αυτή είναι ήδη εδώ και τέσσερα χρόνια υποψήφια και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίσης, το θέμα της αναγνώρισης του κοσυφοπεδίου για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει άμεσα τη Μακεδονία. Γιατί ανεξάρτητα από την θέση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κοσυφοπέδιο και η οποία μπορεί να είναι δύσκολη για ορισμένε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Παρ' αυτά, πολλές χώρε λοιπόν δέχτηκαν την ανεξαρτησία του κοσφοπεδίου και έχουν ακολουθήσει την γραμμή πλεύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν δεν πρόκειται για το θέμα του Κωσυφοπεδίου, αλλά για τη στάση που θα υιοθετήσει η Μακεδονία έναντι του Κωσυφοπεδίου και η χώρα αυτή χρειάστηκε να κάνει πάρα πολλές προσπάθειες για να ευθυγραμμιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, εν κατακλείδη, η Επιτροπή μας και στη συνέχεια η Ολομέλεια είχαν ήδη εκφέρει γνώμη πέρσι ώστε να γίνουν το ταχύτερο δυνατό οι ενέργειες για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση όπως προτείνω και στην εκθεσή μου που θα έχει σαν αποτέλεσμα μετά από τις εκλογές του Μαρτίου που θα γίνει και ο δεύτερος γύρος στη συνέχεια των προεδρικών εκλογών τον Απρίλιο. Αμέσως μετά τις εκλογές αυτές ελπίζω ότι θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και μέσα στην διάρκεια του 2009 το Συμβούλιο θα λάβει την απόφαση για τις διαπραγματεύσεις αυτές γιατί έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο ήδη και αυτό δεν ήταν θετικό. Αυτά. Αυτά είναι λοιπόν τα βασικά σε σχέση με το ψήφισμά μου και τις τροπολογίες που έχουν τεθεί. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάιερ. Θα ήθελα ε, πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στον σκιώδη των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα κύριε Πρέσβη, ε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη θαυμάσια η εισαγωγή στη σημερινή συζήτηση. Δεύτερον, συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής μας ε, ο κύριος Μάια και η δική μου θέση είναι ότι οι ε, συζητήσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως μετά τις ε, εκλογές. Η δουλειά που έχει γίνει από τη Μακεδονία στο δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά εντυπωσιακή και νομίζω πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε. Κύριε Πρέσβη, έχω τρεις ερωτήσεις να υποβάλω. Η πρώτη ερώτηση αφορά σε αυτό το ε, πρόβλημα του ονόματος ε, της χώρας έχοντας κατά νου την ε, ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολιτικής φύσεως το θέμα, μάλλον ερωτώ. είναι πολιτικό το θέμα, θέμα κριτηρίων της Κοπενχάγης ή είναι ένα διμερές θέμα ένα ε, θέμα που αφορά δύο χώρες. Γενικής φύσεως ε, το θέμα, αλλά εξακολουθεί να εφίσταται. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι το εξής. Εσείς ε, πώς ακριβώς αξιολογείτε την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στη Μακεδονία. Έχουμε ελεύθερα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει ελευθερία τύπου και έκφραση των μέσων ενημέρωσης στη Μακεδονία ή όχι. Και τρίτη ερώτηση. Εσείς τι πιστεύετε για τη συγκατοίκηση με την αλβανική κοινότητα στη Μακεδονία, κυρίως μετά την ανεξαρτησία του Κοσφοπεδίου. Η ανεξαρτησία του Κοσφοπεδίου είχε θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες, δηλαδή καμία επίπτωση στο θέμα της Μακεδονίας. Η κυρία της μακεδονιας η κυρια Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μέιερ για την παρουσίασή του. Έχω την αίσθηση ότι η παρουσίαση αυτή ήταν μια πληρέστατη, μας έδωσε μια πληρέστατη εικόνα της κατάστασης και εγώ πιστεύω ότι το θέμα του κοσοπεδίου ε, πρέπει να το εξετάζουμε ξεχωριστά από το θέμα της Μακεδονίας. Εδώ μιλάμε για τη Μακεδονία και μιλάμε και για τη Σερβία και τις προτερότητες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Εγώ λοιπόν υποστηρίζω την άποψή σας ότι κάθε μία από αυτές τις χώρες ε, πρέπει να κρίνεται ανάλογα με τα δικά της τα επιτεύγματα όσον αφορά το ενδεχόμενο έναρξης ε, διαπραγματεύσεων στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν. Έχουμε χάσει πολύ χρόνο και ευθύς ε, εξ αρχής ε, είχαμε μια κατάσταση όπου η Μακεδονία πήρε πολύ νωρίς συμφωνία σύνδεσης και πήρε επίσης πολύ νωρίς ε, την ε, ονομασία της υποψήφιας χώρας, ενώ οι άλλες χώρες ακολούθησαν αργότερα. Όλο και περισσότερες ε, χώρες ζητούν να γίνουν υποψήφιες χώρες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μερικές ελπίζουν να ξεκινήσουν σύντομα διαπραγματεύσεις. Η Μακεδονία βρίσκεται σε αυτή τη θέση εδώ και αρκετό καιρό. Το πρόβλημα με τη Μακεδονία είναι ότι οι διαπραγματεύσεις ε, ε, θα μπορούσαν ήδη να έχουν αρχίσει, αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα με την ονομασία. Μερικοί ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε όμως ε, η κατάσταση να επιδεινωθεί περαιτέρω γιατί ε, και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, πολιτικών ομάδων δεν είναι ενιαία. Εγώ λοιπόν εύχομαι η κατάσταση αυτή να ρυθμιστεί το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και μετά από τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη του ε, συμβασμού διαπιστώνουμε ότι κάποιες πολιτικές ομάδες ανθίστανται, διαφωνούν. Ε, θέλω όμως ε, να πιστεύω ότι τουλάχιστον εδώ στην Επιτροπή μας θα συμφωνήσουμε όλοι και θα στηρίξουμε αυτή τη συμβαστική πρόταση. Και μία ερώτηση προς εσάς. Ποια είναι η δική σας η άποψη Ποια θα ήταν μια ρεαλιστική προσέγγιση, έχοντας βέβαια κατά νου το ότι η Μακεδονία ε, επιθυμεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, από πλευράς χρονοδιαγράμματος. Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει για τη Μακεδονία σε σύγκριση με άλλες χώρες. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε να ε, υπάρχει ταχύτατη πρόοδος. Κύριε Μπέρεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι είναι καλό να ακούει κανείς ε, και από τους δύο ότι η Μακεδονία παρότι τα πράγματα δεν πήγαν και πολύ καλά καταβάλει προσπάθειες να κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός. Έτσι λοιπόν η δική μου η πολιτική ομάδα ελπίζει ότι τώρα πλέον θα μπορέσουμε να λάβουμε ε, υπεύθυνε αποφάσεις. Γνωρίζετε ότι το θέμα της ε, διαφωνίας για την ονομασία εξακολουθεί να παίζει ρόλο. Η δική μου η πολιτική ομάδα ε, κατέθεσε μια τροπολογία που κατατείνει στο ότι θα πρέπει πάρα αυτά να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Μακεδονία. Ήδη τώρα με την ε, αρχή του καινούριου χρόνου υπάρχουν ε, βέβαια συμβαστικές προτάσεις, υπάρχει η πρόταση των σοσιαλιστών που αναφέρθηκε προηγουμένως, δηλαδή αμέσως μετά τις εκλογές του Μαρτίου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Εγώ θα μπορούσα να συμφωνήσω με μια τέτοια απόφαση που θα μπορούσε να ληφθεί εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αν τελείωνε αυτό το μπλοκάρισμα που υπάρχει στο θέμα της ονομοσίας. Νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε σήμερα το θέμα αυτό και να ψηφίσουμε. Για μένα λοιπόν, αν τελικά το ε, πολιτικό μήνυμα είναι να ζητήσουμε από την ελληνική πλευρά να άρει το μπλοκάρισμα που υπάρχει, τότε η έναρξη των διαπραγματεύσεων μετά τις εκλογές σημαίνει, θα συνέμενε αυτό, ότι η Μακεδονία θα μπορούσε να ενταχθεί στα 60 γενέθλια του ΝΑΤΟ, στο ΝΑΤΟ Δηλαδή αν ε, δεν υπήρχε το βέτο από πλευρά ελληνική, ο δρόμο θα ήταν ελεύθερο. Εμένα, εκείνο που με ενδιαφέρει είναι ε, κατά πόσον εσείς ε, κύριε Φουρέρε πιστεύετε ότι αυτή η ενδιάμεση συμφωνία του 1995 κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει ή όχι πρόκειται ε, για μια πολιτική συμφωνία που λέει ότι η ονομασία ε, δεν μπορεί να είναι εμπόδιο για την ε, Μακεδονία έτσι ώστε να ξεκινήσει η και κάποια στιγμή να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και ένα άλλο που με απασχολεί είναι το εξής, ε, ότι η συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτή τη χώρα αποτελεί παραβίαση των κανονισμών που εφαρμόζουμε, ε, παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας και του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και αν ισχύουν όλα αυτά, τότε προφανώς θα πρέπει να γίνουν οι συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση και σε ανώτερο επίπεδο. Όχι εδώ, στη δική μας Επιτροπή, σε πολύ ανώτερο επίπεδο, γιατί δεν είναι δυνατόν να δεχόμεθα τέτοιου είδου παραβιάσει. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τι συμβαστικέ μα προτάσει. Θα είχα χαρεί ο ε, εισηγητή να πει κάτι επ' αυτών των ε, συμβαστικών προτάσεων. Έχουμε μία τροπολογία, μία αλλαγή μάλλον ε, σε αυτή τη τροπολογία τη 15η Ιανουαρίου που είχαν συμφωνήσει οι δύο πολιτικέ ομάδε. Και φαντάζομαι να συμφωνήσουν και άλλοι αν παραμείνει αυτή η ε, συμφωνία. Αλλιώς ε, πρέπει να σας πω ότι στο 5 και στο 6, στα σημεία αυτά, το θέμα της ονομασίας ε, καταλαμβάνει υπερβολικό χώρο, περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Αυτό εμάς μας λείπει, αλλά ίσως μπορεί ο εισηγητής να τοποθετηθεί από αυτού. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φουρέρε ίσως ε, μπορεί να τοποθετηθεί επ' αυτών των ερωτήσεων στον πρώτο γύρο των απαντήσεων. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλα τα εκλεκτά μέλη του Κοινοβουλίου για τις ερωτήσεις τις οποίες έθεσαν. Κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις είναι πολύ δύσκολο για μένα να απαντηθούν. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσω και τα δύο καπέλα θα έχω, τα οποία έχω προσπαθώντας να δώσω απαντήσεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ πάντως. Ξεκινώντας με το χρονοδιάγραμμα, για την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων ένταξης. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι τα πράγματα να προχωρήσουν γρήγορα, να προχωρήσουν γρηγορότερα. Τα πράγματα δεν έχουν προχωρήσει όσο γρήγορα θα θέλαμε γιατί η χώρα δεν εξεπλήρωσε τους στόχους τους οποίους αναμέναμε από αυτήν. Ο Επίτροπος Ρεν ήταν ξεκάθαρος το Μάρτιο του 2008 είπε ότι υπάρχουν οκτώ προτεραιότητες με νέα προτεραιότητες μετά από τις καινούριε εκλογές και εφόσον εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις αυτές θα μπορέσω να σας δώσω μια ημερομηνία αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να εκπληρώσουν κάποιες από αυτούς τους στόχους και η πιο σοβαρή αποτυχία ήταν οι τελευταίες εκλογές και η έλλειψη πολιτικού διαλόγου διαρκούς πολιτικού διαλόγου. Παρ' όλα αυτά οι αντιδράσεις της κυβέρνησης μετά από την έκθεση προόδου του μηνός Νοεμβρίου ήταν ενθαρρυντικοί. Το θέμα είναι να παραμείνει στη σωστή τροχιά η κυβέρνηση και να κατανοήσει ότι εφόσον εκπληρώσει τις μεταρρυθμίσεις αυτές η Επιτροπή θα είναι σε θέση να συστήσει ημερομηνία ένταξης, έναρξης διαπραγματεύσεων. Η διαδικασία είναι ετήσια όπως ξέρετε. Η επόμενη έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ακολουθήσει το φθινόπωρο του 2009. Συνεπώς και εφόσον δεχόμαστε ότι, εφόσον δεχθούμε ότι οι εκλογές θα είναι διεθνούς επίπεδου, αποδεκτές και εφόσον όλα τα άλλα κριτήρια ε, εκπληρωθούν έτσι όπως ορίζονται στη Συμφωνία της Εταιρικής Σχέσης, τότε θα έχουμε πλέον επιχειρήματα στην φθινοπορεινή μας ε, ε, έκθεση να συστήσουμε μια ημερομηνία έναυξης διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν αποκλείει βέβαια το Συμβούλιο το Συμβούλιο Υπουργών, το Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων να διαπιστώσει τα βήματα προόδου τα οποία έχουν επιτελεστεί νωρίτερα αν οι εκλογές ας πούμε πάνε πολύ καλά τότε σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε ε, να αναγνωριστεί κάτι τέτοιο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, την κατάλληλη στιγμή, την εύθετη στιγμή. Πάντως για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πράγματα είναι σαφή. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες έτσι ώστε οι στόχοι να επιτευχθούν και αυτά τα επιχειρήματα πλέον θα είναι αρκετά έτσι ώστε να συστήσουμε μία ημερομηνία για την έναρξη των συνομιλιών για την ένταξη. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Εμείς κάθε μήνα στέλνουμε στοιχεία στις Βρυξέλλες και απαιτούνται μήνες από πλευράς Βρυξελών να αξιολογήσουν τα συνολικά βήματα προόδου. Έχουμε επίσης επαφές με τον ΟΑΣΕ, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την κοινωνία των πολιτών. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη και επ' αυτή της βάσεως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει την πρότασή της. Η έκφραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν γίνεται με ένα μαγικό κόλπο σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αν λοιπόν τα πράγματα πάμε καλά και το ελπίζουμε αυτό, τότε το φθινόπωρο θα μπορέσουμε να συστήσουμε και ημερομηνία γύρω τώρα από το θέμα του ονόματος. Το θέμα του ονόματος είναι πάντα ένα μείζον θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μην συγχαίεται το θέμα αυτό με τις μεταρρυθμίσεις. Και ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε μια ιαδήποτε σύσταση στην τελευταία έκθεσή της γύρω από αυτό δεν έχει τίποτα να κάνει με το θέμα του ονόματος αυτό καθεαυτό, αλλά με το ότι η κυβέρνηση απλά δεν είχε εκπληρώσει τα λεγόμενα κριτήρια της Κοπενχάγης και αυτό το διευκρινίσαμε. Ταυτόχρονα και ο Επίτροπος Ρεν και ο Ήπατος εκπρόσωπος κ. Σολάνα είπαν ότι η επίλυση του προβλήματος του ονόματος είναι βασικό στοιχείο της συνολικής διαδικασίας προς την ευρωπαϊκή ένταξη της χώρας. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε δηλαδή και τις δύο πλευρές έτσι ώστε να βρούνε μια αμοιβαία αποδεικτή λύση. Και αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια μιας ατμόσφαιρας γαλήνης, ενός κλίματος ηρεμίας που να ευνοεί τις διαπραγματεύσεις και έχει μεγάλη σημασία η κυβέρνηση στα Σκόπια να μην αναλαμβάνει δράσεις ή αποφάσεις οι οποίες μπορεί να παρερμηνευθούν. Και γι' αυτό λοιπόν ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του κυρίου Νίμιτς θα ξεκινήσει αρχές Φεβρουαρίου. Εμείς ενθαρρύνουμε λοιπόν την κυβέρνηση να συμμετέχει πλήρως στην διαδικασία και να καταλήξουμε σε μία λύση. Μιλάμε για γείτονες, Μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν εφόσον υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα έλεγα να δώσει ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση. Για τα υπόλοιπα θέματα, τα μέσα ενημέρωσης, όπως διευκρινίστηκε στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το θέμα των μέσων ενημέρωσης είναι προβληματικό πάρα πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί ανήκουν σε ιδιώτες, κάτι το οποίο δεν είναι κακό βέβαια, αλλά οι ιδιοκτήτες αυτοί έχουν πάρα πολύ στενές πολιτικές σχέσεις και αυτό επηρεάζει σαφέστατα τη συντακτική τους γραμμή. Είναι σαφές λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες από τον Σύλλογο των Δημοσιογράφων σε συνεργασία με τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες έτσι ώστε να υπάρξει κάποιος τρόπος για να μπορέσουν τα μέσα ενημέρωσης να λειτουργήσουν με ανεξάρτητο τρόπο και οι συνθήκες εργασίας για τους δημοσιογράφους να βελτιωθούν και να δοθούν έτσι κίνητρα για ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία καθώς πλησιάζουμε τις εκλογές γιατί θα υπάρξουν θα έλεγα προκλήσεις από διάφορα πολιτικά κόμματα τα οποία θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν τα μέσα ενημέρωσης και αυτό είναι κρίμα γιατί τελικά πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα πετύχει πολλά εφόσον διασφαλίσει ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης για τις διακοινωτικές σχέσεις Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε τη Συμφωνία της Αχρίδας σαν ένα πετυχημένο πρότυπο συμφιλίωσης. Προβλήματα υπάρχουν, ειδικά προβλήματα τα οποία έχουν εμφανιστεί τον τελευταίο καιρό, όπως η τάση για διαχωριστικές γραμμές στην εκπαίδευση, κάποια σχολεία τα οποία οδηγούν σε ένταση των συγκρούσεων θα έλεγα ή των διαφορών μάλλον σε σχολικό επίπεδο. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα προωθώντας και ε, διδακτέα ύλη αλλά και δραστηριότητες εκτός σχολείου έτσι ώστε η πολυκοινοτική κοινωνία να γίνει κατανοητή. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα μετά τις εκλογές. Η ανεξαρτησία του κοσυφοπεδίου βεβαίως και επηρέασε τη χώρα οι εθνοτικά Αλβανοί ήταν ευτυχείς από το συμβάν αυτό και κάποια από τα μέλη επίσης και των εθνοτικά Μακεδόνων λέει ο μιλητής το ίδιο. Ε, τελικά είδαμε ότι η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αναγνώριση δεν ήταν εύκολη γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να διατηρήσει καλές σχέσεις και με την Σερβία και έχω την εντύπωση ότι το θέμα του κοσυφοπεδίου και της αναγνώρισής του είναι κάτι το οποίο προχώρησε και έγινε αντικείμενο διαχείρισης με πολύ ευαίσθητο τρόπο και αντικατοπτρίζει την εικόνα και επιθυμία της κυβέρνησης να προωθήσει την περιφερειακή σταθερότητα. Ξέρετε επίσης ότι συμμετέχει και στη Στρατιωτική Επιτροπή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην Βοσνία Ευζεγοβίνη γιατί κάτι το οποίο κόστησε ιδιαίτερα στη μικρή αυτή χώρα γιατί έχασαν 11 στρατιώτες σε ένα δυστύχημα μετά την πτώση ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου. Ε, Αλλά εν πάση περιπτώσει η συμφωνία της Αχρίδας είναι κάτι το οποίο ε, έχει προχωρήσει αρκετά και θα αντιμετωπιστεί εκ νέου το θέμα μετά τις επερχόμενες εκλογές Τώρα έχουμε μόνο τρία λεπτά και έχω τέσσερις ε, ε, ομιλητές. Γι' αυτό περιοριστείτε παρακαλώ σε ένα λεπτό ο καθένας. Κυριλόφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα σύντομο σχόλιο θα κάνω. Πρώτα απ' όλα νομίζω πρέπει να είμαστε ευγνώμονες ε, στον πρέσβη για αυτή την ιδιαίτερα ρεαλιστική προσέγγιση. Επίσης να σας πω ότι εγώ ε, συμμετείχα στην Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή και όλα αυτά που μας είπε ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Όσον αφορά τώρα το πρόβλημα με τα μέσα ενημέρωσης, νομίζω ότι οι ε, περισσότεροι συνάδελφοί μας θα συμφωνούν ότι πρέπει η Μακεδονία να προχωρήσει, να συνεχιστεί η διαδικασία και αυτό που είναι πολύ σημαντικό όπως είπε και ο πρέσβης είναι ότι χρειαζόμαστε τώρα στις επόμενες εκλογές ουσιαστική πρόοδο. Πάντως ε, υπάρχει ένα θέμα ε, για τα μέσα ενημέρωσης που υπήρχε στο τελευταίο μας ε, ψήφισμα και από αυτού δεν υπάρχει πρόοδος. Αναφέρομαι στις ε, ε, στην έλλειψη ανεκτικότητας ε, και στις ομιλίες που υποδαβλίζουν το μίσος. Κοιτάξτε, υπάρχουν τέτοιου είδου περιπτώσει ομιλιών που απευθύνονται σε μια γειτονική χώρα. Και αυτό, αν κάποιοι ισχυριστούν ότι προκύπτει γιατί υπάρχει το πρόβλημα τη ονομασία με την Ελλάδα, κοιτάξτε, δεν είναι αλήθεια, γιατί απευθύνονται και στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία δεν έχει πρόβλημα ονομασία. Θα ήθελα λοιπόν κύριε Πρόεδρε να αναφέρω ένα παράδειγμα του τι ακριβώς συνέβη στα μέσα ενημέρωση σε σχέση με τη Βουλγαρία. Κατά την τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού, μία από τις ε, μεγαλύτερες εφημερίδες της χώρας ε, μας υπενθύμησε για άλλη μια φορά ότι η Βουλγαρία, το κράτος, ε, ε, η κυβέρνηση, όλοι οι Βούλγαροι είναι πρωτόγονοι, ανεκπαίδευτοι και θα παραμείνουν αυτά τα μαύρα βουλγαρικά τέρατα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά τέτοια παραδείγματα και διαρωτώ με γιατί δεν υπάρχει πρόοδο σε αυτό το θέμα. Εγώ μην ξεχνάτε στήριξα και το θέμα τη χορήγης θεωρήσεων γιατί πιστεύω ότι οι μακεδόνε πολίτε ε, θα πρέπει να μπορούν ελεύθερα να ταξιδεύουν στις όμορφε χώρε για να διευθυνθούν και μόνοι ότι δεν υπάρχουν τέρατα στη γειτονιά. Ο κύριο Κυρίτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρεσβευτή για την πλήρη παρουσίαση που μα έχει κάνει, τη κατάσταση που επικρατεί στην πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και επίση σε ό,τι αφορά τις προοπτικές για τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω ένα ερώτημα να σας θέσω. Με ενδιαφέρει να γνωρίσω το κατά πόσο οι εθνοτικές μειονότητες εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο της ε, Μακεδονίας, η βουλγαρική, η σερβική, η αλβανική μειονότητα και όλα αυτά. Ρουμανική συγγνώμη ενότητα. Ο κύριος Στογιάννοφ. σήμερα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να προσθέσω και κάτι σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κυρίλοφ. Εγώ κατέθεσα τρεις τροπολογίες, δύο από τις οποίες ε, είναι φανερό ότι έχουν απορριφθεί από τον εισηγητή Η μία από αυτές αφορά την βία, τη σωματική βία που έχει ασκηθεί κατά των Μακεδόνων οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Βούλγαροι. Θεωρεί ο εισηγητής ότι είναι απαραδεκτή αυτή η βία για τα άτομα αυτά ή είναι και γι' αυτό είναι εναντίον της τροπολογίας μου. Δεύτερο ερώτημα. Έχετε κάποιες πληροφορίες σε σχέση με τις διακρίσεις που ασκούνται εναντίον των ατόμων που έχουν μια βουλγαρική εθνοτική ταυτότητα. Το θέμα της ύπαρξης μιας βουλγαρικής ταυτότητας στη Μακεδονία είναι κάτι το οποίο είναι πολύ παλιό, δεν θέλω να επισέλθω σε αυτό, αλλά υπάρχει μια οργάνωση βουλγαρική στη Μακεδονία που έχει μια ε, υπόθεση που εκκρεμεί στα δικαστήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Κοπά. Πρόεδρε, ε, νομίζω από τη συζήτησή μας φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγχυση το ε, κείμενο της επιτροπής οι δηλώσεις του όλι Ρεν αλλά και η τοποθέτηση του κύρου πρέσβη δείχνουν καθαρά ότι η μη ε, έναρξη των διαπραγματεύσεων οφείλεται στο ότι δεν τηρήθηκαν τα benchmarks που είχαν τεθεί από την ευρωπαϊκή ένωση. αντίθετα όπως προκύπτει μέσα από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν φαίνεται το κλίμα μες στην επιτροπή να είναι ότι βασικός υπέτειος για αυτή την καθυστέρηση είναι το πρόβλημα του ονόματος με την ελλάδα. θέλω μόνο να πω ότι η δαιμονοποίηση ενός κράτους μέλους δεν βοηθάει ε, για όλα τα δεινά τη χώρας δεν βοηθάει να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα δεν βοηθάει να βρεθεί λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τις δύο χώρες για πολύ καιρό και νομίζω ότι είναι σαφές ότι η ελλάδα περισσότερο από άλλες χώρες που είναι πολύ πιο μακριά θέλει μια δημοκρατική χώρα χωρίς εθνικισμούς επειδή ακριβώς γειτονεύει μαζί της είμαστε γείτονες. από την άλλη πρέπει το κοινοβούλιο να μπορέσει να βρει τον τρόπο ώστε να μπορέσει να ε, οδηγηθεί σε λύση και να βοηθηθεί η χώρα να πλησιάσει την ευρωπαϊκή ένωση. Ευχαριστώ. Τώρα λοιπόν ε, θα ακούσουμε τον κύριο Πρέσβη και μετά θα ακούσουμε και σύντομες ε, τοποθετήσεις από τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη αν δεν θα προλάβω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Θα το ήθελα. Ξέρω ότι δεν μπόρεσα να καλύψω όλα τα ερωτήματα του κυρίου Μέγερ. Σε ό,τι αφορά τις μειονοτικές κοινότητες στην ε, Μακεδονία. Υπάρχουν ορισμένε οι οποίε εκπροσωπούνται στο τοπικό κοινοβούλιο. Είναι η μόνη χώρα όπου υπάρχει ένα δήμος του οποίου ο δήμαρχος ανήκει στην κοινότητα των Ρώμα. Πολλά έχουν γίνει λοιπόν για αυτές τις κοινότητες και πρέπει, θα πρέπει να εξάρουμε τις προσπάθειες της μακεδονικής κυβέρνησης στον τομέα αυτό. Αν τώρα υπάρχουν προβλήματα, παραδείγματο χάρη με τη Βουλγαρία, ο καλύτερος τρόπος να επιληθούν αυτά τα προβλήματα είναι με το διάλογο. Όταν υπάρχουν λοιπόν τέτοια προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διάλογο και φυσικά μπορεί κανείς να έχει και πρόσβαση στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, το οποίο μπορεί να επιλύσει ενδεχομένως τέτοια θέματα, αλλά πιστεύω ότι με καλή θέληση και από τις δύο πλευρές θα πρέπει να είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία συνέβησαν στο παρελθόν σε ό,τι αφορά την αναμόχλευση των παθών και την ε, ε την δημιουργία ενό κλίματος μίσους. Νομίζω ότι επίσης η Συμφωνία της Αχρίδας είναι το καλύτερο υπόδειγμα για συμφιλίωση και την οικοδόμηση μιας πολυεθνοτική κοινωνίας η οποία ανταποκρίνεται προς τα συμφέροντα της χώρας αυτής. Και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι είναι πράγματι πεπισμένοι και αποφασισμένοι οι πολίτες της χώρας αυτής να προχωρήσουν να επιτύχουν συμβιβαστικές λύσεις για τα θέματα αυτά, να ξεπεράσουν τα προβλήματα που έχουν με τους γείτονέ τους για να προχωρήσουν προς την οδό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να πρόκειται τώρα στους πολιτικούς ηγέτες να ερμηνεύσουν αυτό το πνεύμα συμβιβασμού και ομόνιας ώστε η χώρα αυτή να περάσει στο επόμενο ορόσημο της διαδικασίας ένταξης. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Ο κύριος Μάιερ για ένα σύντομο συμπέρασμα. Δύο ερωτήματα έχω, κύριε Πρόεδρε, τα οποία αφορούσα και εμένα εξάλλου. Από την κυρία Μπέαρ, καταρχήν, είπε ότι πρέπει να δώσουμε λιγότερη σημασία στο θέμα του ονόματος και των σχέσεων με την Ελλάδα. Μπορώ να καταλάβω τη θέση της. Πριν από ένα χρόνο είχα πει ότι ήταν η ελπίδα μου στο επόμενο ψήφισμα μετά από ένα χρόνο να μην χρειάζεται να θίξουμε καθόλου αυτό το θέμα παρά μόνο να πούμε ότι είχε ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό και ότι επικρατούσαν καλές και θετικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών χάρη σε μια αμεβαία κατανόηση που θα προωθούσε και τη διαδικασία ένταξης. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν έχει συμβεί. Και το αποτέλεσμα λοιπόν των διαπραγματεύσεων για τις τροπολογίες συμβασμού είναι ότι θα πρέπει να πούμε κάτι. Δυστυχώς δεν μπορώ να ικανοποιήσω την κυρία Μπέα, συμφωνώ λοιπόν στην ουσία μαζί της, αλλά όχι στα συγκεκριμένα. Αυτά που ο κύριο Στόιανοφ για τη βουλγαρική μειονότητα. Ο εκφοβισμό και η βία είναι κάτι που καταδικάζω απεριφράστο. Και σύμφωνα με τον κύριο Στόιανοφ πρέπει να τα καταδικάσουμε αυτά τα φαινόμενα. Αλλά υπάρχει και μια άλλη συζήτηση που διατρέχει αυτό το πρόβλημα, που είναι το πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό για του Βούλγαρου. Το ερώτημα έχει τεθεί αν οι Μακεδόνε είναι Βούλγαροι και αν η μακεδονική γλώσσα είναι απλώ μια παραλλαγή τη Βουλγαρική η πλειοψηφία του λαού της Μακεδονίας θεωρεί ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πράξουμε κάτι το οποίο θα θίξει τις ευαισθησίες σε σχέση με το θέμα αυτό. Γι' αυτό εγώ καταδικάζω τη βία και τον εκφοβισμό, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε παράλληλα οποιασδήποτε ενέργειες οι οποίες θα ανατρέψουν τις λεπτές ισορροπίες. Πολλοί Μακεδόνες νιώθουν κοντά στη Βουλγαρία, αλλά όχι τμήμα της Βουλγαρίας. Αυτό δεν πρέπει να το θίξουμε. Ευχαριστώ. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι την Τετάρτη θα ψηφίσουμε. Έχουμε ακόμα χρόνο να ξεπεράσουμε κάποιες διαφορές μεταξύ μας. Κύριε Πρέσβη, και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μας δώσατε για τις ειλικρινείς απαντήσεις σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο δύσκολο σας έργο και φυσικά καλή τύχη για τη χώρα την οποία εσείς, για την οποία εσείς είσαστε υπεύθυνος. Uh, Αγαπητά μέλη της Επιτροπής μας, κυρίες και κύριοι, προχωρούμε τώρα με την συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, με την μονογραφική αυτή συνεδρίαση που αφορά τα θέματα ασφάλειας ενέργειας. Ένας από τους λόγους είναι ότι η Επιτροπή μας έχει διαδραματίσει ένα προεξάρχοντα ρόλο για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας ενέργειας το 2007 και από τότε είναι πάρα πολύ ενεργή για να προσπαθήσει να υπογραμμίσει τη σημασία των προβλημάτων αυτών και να μεσολαβήσει τη διένεξη Ρωσίας-Ουκρανίας. Και έχουμε μια πολύ ενεργή στάση στα θέματα αυτά. Έχουμε ζητήσει να γίνουν μελέτες, να μας δοθούν εμπειρογνωμοσύνες για τα θέματα αυτά Ξέρω ότι υπήρξε η συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Δεν έχει ξεκινήσει η παράδοση αερίου. Αλλά αυτά είναι η κατάσταση την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Κάποια μέρα θα έρθει και το φυσικό αέριο. Και γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε την ασφάλεια φοδιασμού. όχι μόνο στο φως των προηγουμένων καταστάσεων που πήρανε ανησυχητική τροπή λόγω της ασυνέχειας στην παράδοση φυσικού αερίου, αλλά να δούμε και τι θα γίνει και στο μέλλον. Έχουμε λοιπόν ορισμένα πολύ σημαντικά θέματα. Το θέμα της διαφοροποίησης της ε, τροφοδοσίας ενέργεια. Ξέρουμε και πιστεύουμε ότι δεν είναι πια μονάχα ένα πρόβλημα ενεργειακής πολιτικής ή ένα εμπορικό θέμα, αλλά ένα θέμα μέτρων εξωτερικής ε, πολιτικής και προσέγγισης εξωτερικής πολιτικής. Αυτή ήταν και η θέση της Επιτροπής μας στο παρελθόν και η ροή των γεγονότων κατέδειξε την σοφροσύνη μας και το γεγονός ότι είχαμε δίκιο. Έχουμε ζητήσει να γίνουν τρεις, να συνταχθούν τρεις εκθέσεις. Η πρώτη από ένα εμπειρογνώμονα τον καθηγητή Άλαν Ρίλεϊ που είναι καθηγητής δικαίου στο Πανεπιστήμιο του City του Λονδίνου και είναι επίσης και στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Βρυξέλλες και έχει κάνει μια μελέτη για το θέμα του South Stream και του Ναμπούκου. Η προηγούμενη του εμπειρογνωμοσύνη ήταν για το North Stream. Έχουμε και τον Ανδρέα Μόναχαν από το αμυντικό κολέγιο του ΝΑΤΟ στη Ρώμη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ενεργειακό εξωτερικό τομέα θα μας παρουσιάσει τις κύριες κατευθύνσεις αυτής της εκθέσεως η οποία ε, ενεκρίθη σχεδόν ομόφωνα πριν από ένα χρόνο από το Κοινοβουλίο μας και προτείνει περαιτέρω ενέργειες, δηλαδή θα κάνει ένα απολογισμό του τι έχει γίνει και το τι δεν έχει γίνει. Εγώ πιστεύω ότι αν είχαν ληφθεί υπόψη όλες οι συστάσεις της έκθεσής του και είχαν εφαρμοστεί, δεν θα είχαμε αυτή την μεγάλη ενεργειακή κρίση που γνωρίσαμε ή που ακόμα γνωρίζουμε ενδεχομένω, ποιος ξέρει. Και υπάρχει και η τρίτη μελέτη η οποία είχε ζητηθεί αλλά δεν είναι παρόν ο συντάκτης της. Τα θέματα της ε, ασφάλειας του South Stream από την κυρία Ζέινο Μπαράν η οποία ήταν ε, εμπειρογνώμων και στην ακρόαση που κάναμε πριν από 1,5 χρόνο. Θα βρείτε λοιπόν και τις τρεις εκθέσεις στους φακέλους σας και επίσης στο διαδίκτυο στην σελίδα της Επιτροπής μας και έχουμε και τον κύριο Γκέρχαρτ Σαμπατήλ ο οποίος είναι διευθυντής στην ε, Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων στην Κομισιόν και ο οποίος ε, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα στην ε, Γενική Διεύθυνση Ρέλεξη για τα θέματα ασφάλειας ενεργειακής τροφοδοσίας. Έχουμε επίσης και τον νεοστή διοριστέντα εκπρόσωπο του υψηλού εκπροσώπου του κυρίου Σολάνα, τον κύριο Στίβεν Evans. Evans. Και θα αρχίσουμε με τις εμπειρογνώμονες με τη σειρά που την έχουμε αναφέρει. Θα δώσω λόγο στον κύριο Άλαν Ρίλεϊ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαι εδώ, ονομάζομαι Ράιλι και σας παρουσιάζω μια πρώτη παρουσίαση της ε, έκθεσής μου. Θα λάβω υπόψη τα σχόλιά σας και θα προχωρήσω στην τελική μου έκθεση. Δύο, βασικές ε, δύο βασικά θέματα, το ένα το Ναμπούκο και το άλλο το South Stream. Να μιλήσω για λίγα από τα προβλήματα του Ναμπούκο και μετά να περάσω μέσα στο δεκάλεπτο το οποίο έχω στα υπόλοιπα θέματα, οφείλω να είμαι ιδιαίτερο συνθετικός. Το σχέδιο South Stream, το οποίο περιλαμβάνει την οικοδόμη την δημιουργία ενός αγωγού στις νότιες θάλασσες, έχει σαν στόχο την παροχή αερίου στη Νότια Ευρώπη. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι αμφισβητούμενο από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως. Η δυσκολία του South Stream είναι η εξής. Πρώτον, το κόστος της. Μιλάμε για ένα αγωγό, ενός αγωγού, ο οποίος έχει 900 χιλιόμετρα, 900 χιλιόμετρα μήκος, σε βάθος 2.000 χιλιόμετρων κατά τη διάρκεια της διαδρομής την οποία αντίθετα με το North Stream το οποίο είναι σε βάθος μόνο 200 μέτρων και όχι 2.000 μέτρων. Το κόστος είναι υψηλότατο και οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας είναι γύρω στα 20 δις. Μιλάμε για ένα δηλαδή κόστος πάρα πολύ υψηλό και υπάρχουν ιδιαίτερα δύσκολα ερωτηματικά σχετικά με την ικανότητα της Gazprom να χρηματοδοτήσει αυτήν την, αυτό τον αγωγό. Υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο είναι κάτι το οποίο οι βουλευτές σε μια χρονιά εκλογών θα λάβουν υπόψη τους. Μιλάμε για υψηλό κόστος αγωγού, δηλαδή για υψηλό κόστος φυσικού αερίου. Οι Ρώσοι λένε ότι εμείς θα δημιουργήσουμε αυτό το πολύ ακριβό αγωγό και οι καταναλωτές θα πληρώνουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές για το αέριό μας. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από πλευρά σας. Αυτό το οποίο θα έλεγα επιβαρύνει την κατάσταση είναι ότι δεν ε, παίρνουμε επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου. Αυτό το οποίο μας προσφέρουν είναι στην ουσία μια απόκληση από τα σχέδια τα οποία υπάρχουν. Αντί να βάζουν το αέριο ε, στα ουκρανικά δίκτυα τα οποία έχουν ε, θα έλεγα αποσβεστεί δημιουργούμε ένα νέο αγωγό. Το μόνο που κάνει για τον Ευρωπαίο καταναλωτή είναι το να αυξάνει το κόστος. Η ρωσική απάντηση είναι ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα με την Ουκρανία και τα είδαμε και πρόσφατα. Η απάντησή μου σε αυτά που ισχυρίζονται οι Ρώσοι είναι ότι κάνουν την πολιτική επιλογή. Υπάρχει μια πιο φθηνή επιλογή η διαπραγμάτευση ενός καθεστώτος διεθνούς διαμετακόμισης του αερίου μέσω της Ουκρανίας και να υπάρξει δηλαδή ε, ένα καθεστώς ελεγχόμενο ε, μέσω της Ουκρανίας, κάτι το οποίο δεν θα επιβαρύνει τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Γιατί το κόστος ε, του προτινόμενου αγωγού είναι ιδιαίτερο υψηλό. Κάποια άλλα θέματα σχετικά με το South Stream. Για να κατασκευαστεί θα πρέπει να περάσει από οικονομικές ζώνες ουκρανικές ε, και ρουμανικές. Και οι δύο αυτές χώρες θα αξιολογήσουν προσεκτικά το σχέδιο. Η Ουκρανία προφανώς και έχει ένα κίνητρο να είναι κατά του αγωγού λόγω ακριβώς της απώλειας ποσοτήτων από την ίδια της τη χώρα. Η Ρουμανία τώρα αν κατασκευαστεί το αέριο θα κοστίζει πολύ. Το θέλει αυτό το η Ρουμανία. Νομίζω ότι το κόστος δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα προκαλέσει καθυστερήσεις από πλευράς και της Ρουμανίας. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τον Ευρωπαίο καταναλωτή σε σχέση με το κόστος ε, του φυσικού αερίου που θα μεταφέρεται και με την προστιθέμενη αξία. Για τον Αμπούκο τώρα. Το βασικό πρόβλημα είναι από πού θα έρθει το φυσικό αέριο. Ε, εν μία βασική πηγή είναι το Ιράν. Ξέρουμε τι δυσκολίες παρουσιάζει αυτό. Έχουν υπάρξει ε, πάρα πολλές ε, αυξήσεις στην εσωτερική ζήτηση. Έχει υπάρξει πλήρης απουσία επενδύσεων στην ε, παραγωγή αερίου στο Ιράν και παρότι έχει τρίτο μεγαλύτερο απόθεμα το Ιράν εισάγει αέριο και επιπλέον υπάρχουν και οι κυρώσεις εις βάρος του Ιράν κάτι το οποίο δημιουργεί την εξαγωγή αυτή δύσκολη. Υπάρχει δυναμικό βέβαια ακόμα και αν αναιρεθούν οι περιορισμοί οι εμπορικοί σήμερα το, θα πρέπει να υπάρξουν τεράστιες επενδύσεις για να αυξηθεί η παραγωγή και με το Ιράν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε σύνδεση επίσης και με τον αραβικό αγωγό. Εδώ έχουμε θέματα ασφαλείας τα οποία δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Το Τουρκμενιστάν είναι κάτι το οποίο προσφέρεται περισσότερα από τις δύο περισσότερες πηγές κάποιες ε, μορφές ελέγχου πρόσφατες δείχνουν ότι το Τουρκμενιστάν έχει ε, κοιτάσματα. Το θέμα είναι θέμα κόστους, είναι θέμα χρόνου και αυτό θα δημιουργήσει αύξηση στις τιμές. Ε, υπάρχει επίσης και η δυνατότητα της κυβέρνησης να καλύψει τις ανάγκες που έχει η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, κάτι το οποίο λειτουργεί πολλές φορές ανταγωνιστικά και δυστυχώς ε, η πρόταση για τον κοινό αγωγό μέσω της Κασπίας από ό,τι φαίνεται λόγω της ρωσικής τάσης δεν προχωρά. Πάντως η πιο ε, καλή πιθανότητα είναι από το Αζερμπαϊτζάν. Εκεί υπάρχουν τεράστιες ποσότητες αερίου, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όμως ότι το Αζερμπαϊτζάν θα πρέπει να βγάζει αέριο αλλά να περνάει από τη Γεωργία και την Τουρκία, κάτι το οποίο δημιουργεί και αυτό κόστος. Υπάρχει λοιπόν αέριο αλλά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για την μεταφορά του στη Δυτική Ευρώπη. Έχουμε προβλήματα επίσης και για τον ρόλο της Τουρκίας στην παράδοση του αερίου η Τουρκία θέλει ένα μεγάλο κομμάτι, έχει και προβλήματα σε σχέση με τις διαδικασίες διαμετακόμισης και το θέμα είναι πόσο γρήγορα μπορεί να προχωρήσει ε, το σχέδιο αυτό λόγω της αυξανόμενης τουρκικής ζήτησης. Ένα άλλο θέμα είναι η χρηματοδότηση του Ναμπούκο. Η οικονομική κρίση δεν βοηθάει καθόλου. Υπάρχει ανάγκη να δοθούν ε, εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση πριν ξεκινήσει το Ναμπούκο. Αν οι στόχοι στον τομέα της ασφάλειας τους οποίους έχουμε παίζουν ρόλο, το θέμα είναι πώς θα συνδυάσουμε τις οικονομικές δυνατότητες που έχουμε για να προχωρήσει το Ναμπούκο. Αυτό θα πρέπει να γίνει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, συνειδητοποιώντας ότι πρώτον θα καθυστερήσει το σχέδιο αυτό και σε λίγο καιρό το Ναμπούκο, για λίγο καιρό το Ναμπούκο δεν θα μπορεί να λειτουργεί ε, ε, με πλήρη δυνατότητα μεταφοράς και το θέμα της μεταφοράς του αερίου της Κεντρικής Ασίας στην Ευρώπη είναι κάτι το οποίο δεν έχει ε, βρει τη λύση η οποία αξίζει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το South Stream δεν είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη θα πρέπει να αποφύγει να έρθει ε, στην κατάσταση να χρηματοδοτήσει ένα αναγωγό ο οποίος θα κοστίζει πολύ και δεν δίνει επιπλέον ποσότητες. Απαιτείται να βρεθεί ένα πρωτόκολλο διαμετακόμισης μέσω της Ουκρανίας. Τώρα για τον Αμπούκο το θέμα είναι ότι υπάρχει αέριο, υπάρχουν πηγές αερίου, υπάρχουν όμως ερωτηματικά για το αν η Ευρώπη θα βοηθήσει την διασφάλιση της προμήθειάς της σε ενέργεια. Υπάρχει θέμα ασφαλείας δηλαδή από τη μία και υπάρχει και θέμα κόστους και από την άλλη. Λοιπόν, τώρα για το υγροποιημένο αέριο είναι μια επιλογή η οποία θα πρέπει να εξεταστεί. Μπορεί να προεκταθεί ο αγωγός Μπακού Τουρκίας που πηγαίνει στον λιμένα τον τουρκικό του Τσεχάν και από εκεί μπορεί να έρχεται με σκάφη, με πλοία. Αυτό είναι κάτι το οποίο κοστίζει, όχι ε, κοστίζει όσο ο νέος αγωγός South Stream, αλλά σίγουρα είναι μια δυνατότητα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων που είναι διαθέσιμα και σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο. Και επίσης υπάρχει και το λεγόμενο Nabucco Light, έτσι το ονομάζω, δηλαδή υπάρχει ο, η σύνδεση Τουρκίας-Ελλάδας και ένα τμήμα του αερίου μέσω της Τουρκίας έρχεται στην Ελλάδα. Το θέμα είναι μπορούμε να δημιουργήσουμε την γραμμή από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία. Μπορούμε να ενισχύσουμε τον αγωγό Τουρκίας-Ελλάδας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βάση πάση περιπτώσει τους υπάρχοντες αγωγούς στην Νότια Ευρώπη και να ακολουθήσουμε μια, μια στρατηγική light για τον Αμπούκο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλά οικονομικό σαν θέμα, αφορά και την ίδια την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό πρέπει να εξετάσουμε αν υπάρχει πολιτική βούληση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να πάει σε σχέση με τον Αμπούκο και τις συνέπειες που θα δημιουργήσει. Θέλει τον Αμπούκο Light, θέλει κάποια άλλη λύση, πρέπει να εξετάσει τις συνέπειες σε επίπεδο ασφαλείας. Νομίζω ότι δεν μπορώ να ξεπεράσω τα 10 λεπτά μου ακόμα και αν είμαι πανεπιστημιακός. Ευχαριστώ κύριε Ράιλι. Και τώρα έχουμε το λόγο, έχει ο Andrew Monaghan από το αμυντικό ε, κολέγιο, από την από την υπηρεσία του ΝΑΤΟ στη Ρώμη. Ε, κυρίες και κύριοι, μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να λάβω το λόγο και που μπορώ να αναφερθώ σε δύο έγγραφα τα οποία μου άρεσε πάρα πολύ να τα διαβάσω. Ε, όπως και ο παρακαθήμενός μου και εγώ έχω δέκα λεπτά για να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο βέβαια είναι τεράστιο. Θα προσπαθήσω να εστιάσω την προσοχή μου σε δύο-τρία θέματα για να προκαλέσω τη, τις ερωτήσεις και να δώσουμε τις ε, δέουσες απαντήσεις. Το βασικό θέμα που θέλω να θίξω είναι ότι από όποια πλευρά και αν το δούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξτάσει το θέμα της ε, ενέργειας, της ασφάλειας ενέργειας, έχοντας κατά νου και τις προκλήσεις, την ασφάλεια και βεβαίως και το οικονομικό θέμα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε εκτεταμένη οικονομική ύφεση. Θα έχουμε να ανταγωνιστούμε παίκτες που δεν ακολουθούν τους ίδιους κανόνες και σε τελική ανάλυση μιλάμε και για ενεργειακή ανασφάλεια. οι εκθέσεις εστίασαν την προσοχή τους στο να εξετάσουν εν μέρη εσωτερικά θέματα για να υπάρχει εσωτερική συνοχή, ε, υποδομή, αλληλεγγύη. Νομίζω ότι αυτά αποτελούν ένα πολύ σημαντικό τμήμα οποιασδήποτε ενεργειακής στρατηγικής. Για μένα λοιπόν αυτό που παίζει ρόλο είναι να αναλάβει κανείς τη στρατηγική πρωτοβουλία. Αν υπάρχει εσωτερική συνοχή, ως Ένωση θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις ε, προκλήσεις και παράλληλα θα μπορέσουμε να αδράξουμε τις ευκαιρίες ε, καθοδόν όπως αυτές προκύπτουν. Για να καταλάβετε ε, τι θέλω να πω, θα ξεκινήσω με τη Ρωσία αυτή είναι το επίκεντρο των σκέψεών μας σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια. Μετά θα αναφερθώ σε δύο άλλα θέματα, στο θέμα της ε, διαφοροποίησης της ενέργειας. Εκεί θα εστιάσω την προσοχή μου σε πηγές και διαδρομές και το κάνω αυτό σκόπιμα γιατί αυτή εξάλλου είναι και μία από τις βασικές προτάσεις που αναφέρονται στην έκθεση. Και τρίτον θα εξετάσω σύντομα το ρόλο του ΝΑΤΟ στην ενεργειακή ασφάλεια ε, ως εκ τούτου θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ε, έρθει σε επαφή με όλους τους ε, εταίρους και με αυτούς που υπάρχουν τώρα και με αυτούς που θα θελήσουμε να έχουμε εφόσον υπάρξει διαφοροποίηση. Υπάρχουν τρία θέματα που αφορούν στην, στη σχέση με τη Ρωσία. Πρώτον, όπως θα γνωρίζετε, η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει αυτές τις σχέσεις για να αποκτήσει πολιτικό βάρος στην Ευρώπη. Δεύτερον, υπάρχουν και γεωλογικοί ε, περιορισμοί όσον αφορά την παραγωγή πετρελαίου και αερίου στη Ρωσία και κατόπιν, όπως γνωρίζετε, η Ρωσία έχει δύσκολες σχέσεις με τους γειτονές της. Εγώ θεωρώ ότι το κλειδί σε όλα αυτά είναι οι περιορισμοί που υπάρχουν στο δυναμικό παραγωγής της Ρωσίας, στην υποδομή της και στις δύσκολες σχέσεις που έχει με τους γειτονές τους. Αυτές είναι οι βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στις σχέσεις της με τη Ρωσία ε, έχουμε και πρέπει να έχουμε κατά νου τις ε, διαφωνίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία αυτή τη στιγμή και πώς αυτές επηρεάζουν την Ευρώπη. Νομίζω ότι ε, σιγά σιγά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσει να αναδύεται μια προοπτική Ρωσίας. Θα έχετε διαβάσει όλοι φαντάζομαι ε, την, ε, τον ανακοινωθέν τύπου 8 Ιανουαρίου του Πρωθυπουργού Πούτιν. που λέει ότι αν θέλετε πρέπει να κάνετε κάτι εγώ νομίζω ότι η Ρωσία θα συμπεριλάβει την ενέργεια στις ε, προτάσεις της ε, αναθεώρησης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Φαντάζομαι πολύ θα γνωρίζετε ότι προτείνουν μια τέτοια ανανέωση του οικοδομήματος ασφάλειας και υποπτεύομαι ότι αυτό ε, θα συνδυαστεί με την αναγκαιότητα να αναθεωρήσουμε και το όλο οικονομικό θέματα δηλαδή ότι πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα της ασφάλειας, το θέμα της ενέργειας και καταλήγουμε στο ότι το ενεργειακό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λειτουργεί και ίσως πρέπει να αναθεωρηθεί. Και βεβαίως μπορεί κανείς να πιστεύει ότι διαφωνεί η ε, Ρωσία με το πρωτόκολλο και τη συμφωνία περί ενέργειας. Όταν έχουμε να κάνουμε τη Ρωσία πρέπει να έχουμε κατά νου και το ότι η Ρωσία θα αντιμετωπίσει σημαντικά οικονομικά προβλήματα κατά το 2009 τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν και σε ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις στη Ρωσία. Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου και πίεση που μπορεί να ασκηθεί ε, στις σχέσεις Gazprom και κράτους. Επιτρέψτε μου να ασχοληθώ λιγάκι με τη διαφοροποίηση στον τομέα της ενέργειας. Βεβαίω καλό είναι αυτό, καταρχήν, εγώ δεν θα το αμφισβητήσω, όμως με τον τρόπο αυτό ε, θίγονται αρκετά θέματα. Πρώτα απ' όλα, η διαφοροποίηση. Πώς μπορεί αυτή να ενισχύσει την αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό αυτό, και διαφοροποιήσουμε περαιτέρω τις πηγές μας, τότε θα ενισχυθεί και το όλο ερώτημα ε, ποια είναι αυτή η ενεργειακή απειλή και απέναντι σε ποιον απευθύνεται. Έτσι κι αλλιώ ε, υπάρχει δυσκολία να έχουμε ενιαία ερμηνεία από αυτού. Και αν υπάρχει διαφοροποίηση θα ενισχυθεί περαιτέρω ο προβληματισμός ε, σε σχέση με αυτό το ερώτημα. Και πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε περαιτέρω διαφοροποίηση χωρίς αλληλεγγύη. Πώς θα συμφωνήσουμε, πού πρέπει να διαφοροποιήσουμε. Τρίτον, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια υποδομή, ποιος θα πληρώσει τελικά για τη διαφοροποίηση της υποδομής, έχοντας κατά νου τις δύσκολες ε, συνθήκες ε, στην οικονομία που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα τρία ερωτήματα που πρέπει να εξετάσουμε και να δώσουμε συνεπέστερες απαντήσεις επ' αυτών. Και κάτι άλλο. Θα πρέπει να διερωτηθούμε ποιες επιπτώσεις θα έχει η διαφοροποίηση στους εταίρους μας. Εάν προσπαθήσουμε να διαφοροποιήσουμε μόνοι μας, χωρίς τους εταίρους, αυτοί τι θα κάνουν, θα αναζητήσουν ε, άλλες ε, σχέσεις προφανώς, δικές τους και με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει περαιτέρω απομάκρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους εταίρους της. Όταν έχουμε κατά νου τη διαφοροποίηση, τότε βεβαίως ο στόχος είναι να έχουμε ως δυνατόν περισσότερες πηγές, ε, διαδρομές και μορφές ενέργειας. Ένα στόχος της διαφοροποίησης, κυρίως στο αέριο, ε, είναι να ξεφύγουμε λιγάκι από τη Ρωσία, που είναι βασικός προμηθευτής, και να αναζητήσουμε άλλους εταίρους ε, που είναι πιο σταθεροί μακροπρόθεσμα. Εδώ ο νότιος διάδρομος προβάλλεται ιδιαίτερα, όμως εγώ διερωτώ πόσο, πόσο προχωράμε με αυτή τη διαφοροποίηση το καλοκαίρι έγινε η συνάντηση κορυφής και προέκυψε ότι ο νότιος διάδρομος είναι περίπλοκος, ασταθής, ε, περιλαμβάνει τον Αγκόνο Καραμπάχ, επίμαχο αυτό, ε, ένταση στις σχέσεις μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι ακόμα και εάν ενισχύσουμε τους ε, αγωγούς BTC, BTE και άλλους αγωγούς στον Κάφκασο, παρόλα αυτά θα υπάρχει απειλή για θέματα ενέργειας και ασφάλειας. Αν πάμε στην Κεντρική Ασία, ε, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε αξιόπιστους εταίρους με αξιόπιστες πηγές. Αυτή η σχέση θα είναι καλύτερη, θα προάγει καλύτερα τα συμφέροντά μας. Σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλά από τα επιχειρήματα υπέρ της διαφοροποίησης ε, είναι λίγο κοντόφθαλμα. Δηλαδή λένε να φύγουμε από τη Ρωσία, αλλά χωρίς να λένε πού να κατευθυνθούμε. Και ε, είμαστε σίγουροι ότι το Τουρκμενιστάν ε, θα είναι πολιτικά πιο αξιόπιστο ή άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, έχουν μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερο δυναμικό παραγωγικότητας ε, και ίσως να είναι και πιο ε, σταθερές πολιτικά από τη Ρωσία. Υπάρχει και αυτό το επιχείρημα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να σκεφτούμε το θέμα διαφορετικότητας. Είπαμε έχουμε τους BTC, BT, το Ναμπούκο. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε κατά ότι δεν ανταλλάσσουμε την Ουκρανία και την, με την Τουρκία να πάμε όλα μας τα αυγά από το ένα καλάθι στο άλλο. Βεβαίως και η Τουρκία είναι καλύτερος εταίρος όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είναι και στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος ε, της Τουρκίας. Ακούσαμε από το καθηγητή Ράλι, υπάρχουν όμως θέματα όπως ε, κατανάλωση αερίου, ε, σχέσεις με τη Ρωσία. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για να διορτηθούμε κατά πόσο πράγματι μπορούμε να έχουμε πραγματική διαφοροποίηση. Ας πάμε πιο κάτω, στη Μέση Ανατολή, ως εναλλακτικό προμηθευτή, ως εναλλακτική περιοχή. Καλό αυτό. Όμως δεν είναι και αυτή ιδιαίτερα σταθερή η περιοχή. Επιπλέον, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση προμηθεύεται το πετρέλαιό της από τη Μέση Ανατολή, έχει νόημα να προμηθεύεται και το αέριο από την περιοχή χωρίς να υπάρχει στρατηγική διαφοροποίηση. Ας πάρουμε τη Βόρεια Αφρική, τη Δυτική Αφρική. Παρεμφερεί σε συνθήκες ισχύουν και εκεί. Θα έλεγα λοιπόν ότι ίσως να αμφισβητούμε τη σταθερότητα κάποιων σημαντικών ε, προμηθευτών αερίου και κάποιων ε, διαδρομών. Γι' αυτό, αν μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι η εμπορική διαφοροποίηση έχει νόημα, θα πρέπει να ε, αμφισβητήσουμε και τα πολιτικά και οικονομικά στοιχεία αυτής της διαφοροποίησης και θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο δεν αναφέρεται άμεσα στην έκθεση, το οποίο αφορά ήδη υπάρχοντες εταίρους. Αναφέρθηκε ο Διεθνής ε, Οργανισμός Ενέργειας. Ε, υπάρχει και η σχέση μας με τον ΝΑΤΟ. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντική αυτή η εταίρεια έχοντας ε, κατά νου την πιθανότητα τρομοκρατικών επιθέσεων, πειρατιών, υπάρχουν αυτά ή ε, συγκρούσεων ε, ε, για το θέμα της παροχής ενέργειας. Ας αναφέρω τώρα κάποια πλονεκτήματα στη σχέση μας με το ΝΑΤΟ. Πρώτα απ' όλα, το ΝΑΤΟ υποστηρίζει ότι έχει περιορισμένο ρόλο και προσπαθεί να συμπληρώνει άλλους σημαντικούς οργανισμούς συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διεκδικεί κυρίαρχο ρόλο και επιφέρει γενικότερα πλεονεκτήματα στην ενεργειακή ασφάλεια. Μετά τον ΝΑΤΟ έχει πολύ περισσότερου εταίρου. Παραδείγματο χάρη συμπεριλαμβάνει και τι ΗΠΑ και τον Καναδά, την Νορβηγία, την Τουρκία, που είναι σημαντικέ χώρε για την ενέργεια. Έχει και μεσογειακού εταίρου στη Μέση Ανατολή, έχει σχέσει και με τη Ρωσία. Έχει λοιπόν ε, πολλούς εταίρους που είναι καθοριστική σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια. Εξάλλου έχει άλλες δυνατότητες διαχειρισμού ε, της ενεργειακής ασφάλειας, άλλους από αυτές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σχέση με την θαλάσσια ασφάλεια ή το υγροποιημένο αέριο. Αν θέλετε, αυτό σε μεγάλο βαθμό μεταφέρεται μέσω θαλάσσης. Άρα παίζει ρόλο εδώ η επαγρύπνηση στη θάλασσα. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχω κι άλλα να πω, αλλά αυτά είναι κάποιες ελλείψεις που υπάρχουν στην έκθεση και πρέπει να τα σκεφτούμε. Να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τους υπάρχοντες ε, τέρους. Ε, και καταλήγω σε ορισμένα συμπεράσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταγωνιστεί για την ενεργειακή της ασφάλεια σε έναν ασταθή κόσμο. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε απαραίτητα εργαλεία. Τα τελευταία δύο χρόνια συμφωνήσαμε για το τι πρέπει να κάνουμε. Όμως πρέπει να προσιλητήσουμε και κράτη που δεν είχαν σκοπό να ενταχθούν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πρέπει να καταφύγουμε στους παλιούς μηχανισμούς της εξωτερικής πολιτική το χρονοδιάγραμμα, τελευταίο μου σχόλιο, ποιο θα πρέπει να είναι περίπου αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι 20, 10, 15 και ούτω καθεξής. Ε, να έχουμε μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με αυτό το χρονοδιάγραμμα. Πώς αυτό θα σχετίζεται με τους δικούς μας τους εταίρους. Ποιο είναι το δικό τους το χρονοδιάγραμμα. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δρομολογήσει μια πολιτική μεταρρυθμίσεων, να εντοπίσει τις αδυναμίες των εταίρων, να προσπαθήσει να δει ε, πού ε, χρειάζονται βοήθεια και όχι ποια είναι τα ατού τους. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζεται σε θέματα ισχύω ε, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο το επιθυμούν οι εταίροι. Και γι' αυτό ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την προσοχή σας και σε ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Ζαμπατήλα από την Γενική Διεύθυνση ΡΕΛΕΞ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με τις δύο αυτές μελέτες και ενδεχομένως υπάρχουν και αντιφατικά στοιχεία στις μελέτες αυτές. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση πάντως λαμβάνει χώρα σε μια στιγμή που είμαστε όλοι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι στο εύθραυστο και στο πόσο τροτό είναι ο εφοδιασμός ενεργείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ένα ερώτημα το οποίο μας απασχολεί όλους και πάρα πολλά από τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί στην ε, συζήτηση που κάναμε τον προηγούμενο Νοέμβριο για τα θέματα ενεργειακής ασφάλειας έχουν γίνει πράγματι πάρα πολύ επίκαιρα. Θέλω τώρα να σταθώ στο γεγονός ότι η ασφάλεια εφοδιασμού στην ενέργεια έχει τρεις πτυχές. Έχει την εξωτερική πτυχή αλλά και την εσωτερική πτυχή, την πτυχή της εσωτερικής αγοράς. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο της εσωτερικής αγοράς να μπορέσουμε να έχουμε μια αλληλεγγύη μεταξύ μας όπως έγινε και τις ε, τελευταίες μέρες. Χρειάζεται αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών αλλά επίσης αυτή η αλληλεγγύη θα πρέπει να υλοποιείται και μέσω διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια σειρά από σχέδια υποδομών τα οποία θα πρέπει να μας συνδέσουν προς την νοτιοανατολική Ευρώπη και προφανώς αυτό προϋποθέτει ότι θα έχουμε μια ενιαία φωνή ως Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντα και αυτό είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η αντιμετώπιση των κρατών μελών για την ενεργειακή ασφάλεια έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση και βέβαια με βάση την ε, κατάσταση που έχουν σε ό,τι αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές φωνές και διαφορετικές προσεγγίσεις. Η πρώτη πτυχή λοιπόν για μένα της ασφάλειας εφοδιασμού είναι η, η εσωτερική πτυχή της εσωτερικής αγοράς. Στη συνέχεια πρέπει να εξετάσουμε και την εξωτερική βέβαια πτυχή. Αυτή είναι μια νέα διάσταση που μας έχει δείξει ότι αυτό το θέμα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παραμελήσουμε και δεν είναι η πρώτη φορά που εμείς αντιμετωπίζουμε προβλήματα εφοδιασμού με το φυσικό αέριο. Και φυσικά υπάρχουν και γι' αυτό κάποιες αιτίε. Οι αιτίε είναι ότι εμείς έχουμε κρατήσει μια στάση η οποία ήταν ίσως αισιόδοξα. Δεν είδε τον αναδυόμενο εθνικισμό σε επίπεδο παραγωγής και ε, χρήσης της ενέργειας σαν ένα όπλο και τις νέες αναδυόμενες γεωγραφικές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο ευρωπαϊκό. Ο νότιος λοιπόν διάβλος ενέργειας είναι ένα από τα έξι κέρια προγράμματα υποδομών τα οποία συζητήσαμε τον προηγούμενο Νοέμβριο και έχουμε τις δύο αυτές εναλλακτικέ λύσεις οι οποίες αναφέρθηκαν. Σίγουρα η διαφορά είναι αυτή η οποία παρουσιάστηκε από τους ομιλητές. Το South Stream είναι ένα σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος, αλλά το Ναμπούκο είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκού συμφέροντος, αν θέλετε, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Και θα πρέπει να λύσουμε όλα τα προβλήματα και τα οποία μας απασχολούν για τα σχέδια αυτά εδώ και πολύ καιρό να τα επιλύσουμε. Το επόμενο βήμα είναι η διάσκεψη η οποία θα γίνει στην ε, Βουδαπέστη για τον, ε, για τον αγωγό του Ναμπούκο και ελπίζω ότι από εκεί θα προκύψουν κάποιες λύσεις και θα μπορέσουμε σύντομα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτών των δύο σχεδίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μέσω αυτών σημαντικά σχέδια τα οποία δεν αφορούν μονάχα την προέλευση του φυσικού αερίου αλλά και την διέλευσή του. Όταν θέλουμε να δούμε τώρα την ενεργειακή πολιτική σαν σύνολο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη το Σεπτέμβριο του 2007 είχε τονίσει στο ψήφισμά του ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα ακόμα για τα θέματα αυτά, εδώ η εσωτερική διάσταση της ενέργειας έχει να κάνει και με το, ενεργεια... με το πακέτο το κλιματικό. Η εξωτερική πτυχή έχει να κάνει επίσης και με τις σχέσεις που έχουμε με τους γείτονέ μας και με τις ε, με τον τρόπο αντιμετώπισή του, όπω δίνει και το παράδειγμα αυτό της πρόσφατης κρίση. Έχουμε την οδηγία για την αποθήκευση φυσικού αερίου, ως ένα παράδειγμα οδού που μπορούμε να ακολουθήσουμε και ίσως θα πρέπει να βρούμε ταχύτερους τρόπους να προχωρήσουμε σχέδια υποδομών, να δώσουμε νέες δυνατότητε χρηματοδότησης, να δώσουμε πολιτική υποστήριξη για τη δημιουργία αυτών των υποδομών, ώστε να πραγματοποιηθούν ταχύτερα. Ίσως θα μπορούσα να κλείσω εδώ κύριε Πρόεδρε. Αν υπάρχουν τώρα κάποια ερωτήματα θα μπορούσα φυσικά να επανέλθω σε πιο ειδικά σημεία. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Σαμπατήλ. Πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θέλω να προσθέσω και εγώ κάτι ακόμα για το Ναμπούκο και το πολιτικό βάρος αυτού του θέματος που μας απασχολεί. Για το Ναμπούκο, εσείς Δόκτωρ Ράιλι δεν εξετάσατε τον ε, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα αποκλείοντας πηγές ε, εφοδιασμού όπως είναι το Ιράν ενώ συγχρόνως υπογραμμίσατε τα όρια του τι μπορεί να προκύψει από τις πηγές της Κασπίας και της Κεντρικής Ασίας. Αν έχουμε μία πολύ αισιόδοξη αντιμετώπιση, ίσως υπερβολικά αισιόδοξη, ότι το πρόβλημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν θα ξεπεραστεί, και θα υπάρξει και εξασφάλιση της σταθερότητας του Ιράκ, κάτι το οποίο είναι αρκετά μακρόπνοο σαν προοπτική, μπορεί κανείς να περιμένει και οι δύο αυτές χώρες να δώσουν φυσικό αέριο για τον Αμπούκο και να καλύψουν τη χωρητικότητά του. Και το λέω αυτό με έναν τρόπο ο οποίο δεν είναι δεσμευτικός βέβαια, χρησιμοποιώντας την ε, δυνατότητα της κοινοβουλευτικής διπλωματίας εγώ είχα έρθει σε επαφή με τον κύριο Τζελίλη, τον υπεύθυνο για την πυρηνική διπλωματία του Ιράν και μίλησα επίσης και με τον κύριο Σαφάρη, τον ε, αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, που μου είπε ότι εάν και ξέρετε βέβαια ποια είναι η πραγματικότητα σε γεωπολιτικό επίπεδο πολλές φορές αλλά αυτή τη στιγμή έχουν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα διαθέσιμα τέσσερα τα έχει ε, ζητήσει η Ελβετία και τα άλλα έξι θα μπορούσαν να γίνουν διαθέσιμα, μέσα σε δύο χρόνια θα μπορούσαν να μας παρέχουν 40 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ενώ ο Ναμπούκο θα μας δίνει 31 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή στην, στον έκτο όροφο μιλάει στη συνέλευση των Προέδρων Πολιτικών Ομάδων ο κύριος Ερντοάν και όταν έχουμε επαφή με πολιτικούς ή κοινοβουλευτικούς από την Τουρκία πάντα τίθεται το θέμα της παροχής φυσικού αερίου γιατί η Τουρκία παίζει ένα κομβικό ρόλο όπως αναφέρθηκε και από τον συναδελφό μας από το αμυντικό κολέγιο του ΝΑΤΟ. Και ο για Χόπτε Σέφερ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ήταν επίσης παρόν και με τον οποίο συναντήθηκε ο κύριος Πέτερν και ο κύριος Φων Βογκάου από την Επιτροπή μας σε σχέση με τα θέματα της ε, ασφάλειας εφοδιασμού για τον ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο θέλω να πω λοιπόν εν κατακλείδη είναι ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες οι οποίες βρίσκονται στο απότερο ίσως μέλλον αλλά οι οποίες θα μπορούσαν πραγματικά να είναι εναλλακτικέ λύσεις. Μιλάμε λοιπόν για διαφορετικές πηγές ε, ε, ενέργειας και διαφορετικούς διάβλους. Γιατί τώρα όλα αυτά είναι τόσο σημαντικά όλο και περισσότερο κατανοούμε ότι αυτά είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλεια και ο κ. Μόναχαν μας το πει βεβαίω ότι πια είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής και πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής. Ακολουθώντας και αυτά τα οποία αναφέρει η ίδια η στρατηγική της Ρωσίας που λέει ότι τα ενεργειακά της προϊόντα θα χρησιμοποιηθούν και για στρατηγικούς λόγους και σκοπούς. Επίσης, η ανασφάλεια στο ενεργειακό τομέα έχει επιπτώσει για εκατομμύρια πολιτών μας και θέτει την βιομηχανία μας σε μια πολύ δύσκολη θέση και εμείς είμαστε εδώ για να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντα των πολιτών. Το πρόβλημα της ανασφάλειας λοιπόν έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πλέον μονάχα σαν ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται σαν ασθενά εμπορικό ή βιομηχανικό θέμα και κλεισμένο το θηρόν. Πλησιάζουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές και σύντομα σε τέσσερι ή σε πέντε μήνες όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υποψήφοι θα πρέπει να είναι υπόλογοι στο, στους εκλογείς τους σε σχέση με αυτά τα οποία έπραξαν για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει η θέρμανση των σπιτιών και των διαμερισμάτων μας για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας μας και οι βιομηχανίες μας. Τι κάνατε λοιπόν θα μας πούν για να μην αντιμετωπίσουμε πάλι την ίδια κρίση που αντιμετωπίσαμε πρόσφατα και τις ακραίες καταστάσεις που έχουμε δει σε χώρες όπως η Βουλγαρία. Και θα τεθεί το ερώτημα αν υπάρχει αρκετή αλληλεγγύη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε ο Διευθυντής ο κ. Σαμπατήλα, έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία, είτε είναι τεχνικά είτε νομικά κτλ. Όλα αυτά καταδεικνύουν την πολιτική σημασία, την εξέχουσα πολιτική σημασία αυτού του πάρα πολύ σημαντικού οριζοντίου θέματος όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε ένα πρωτοπόρο ρόλο επισημένοντας τη σημασία του. Και πράγματι θα πρέπει να κατανοηθεί η σημασία των προσπαθειών μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν αυτό το οποίο ξεκίνησε την προσπάθεια να τονίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή τη διαμάχη ως μπλοκ και έφερε τα άλλα κοινωτικά όργανα στις διαπραγματεύσεις προσκαλώντας την Gazprom και μετά τους ε, ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας στη συνεδρίαση την έκτακτη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Ξεκινώ λοιπόν τη συζήτηση και δίνω το λόγο στον κύριο Πάσκο, ο οποίο είναι αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω ότι αυτά τα οποία συνέβησαν αυτό το χειμώνα μας έπεισαν να εξετάσουμε το πρόβλημα με μεγάλη σοβαρότητα. Την προηγούμενη φορά συζητήσαμε το θέμα αλλά δεν εφαρμόσαμε τα συμπέρασμα στο οποίο είχαμε καταλήξει. Τώρα έχουμε καταλήξει εκ νέου στα ίδια συμπεράσματα. Θα τα ονόμαζα και πιο σημαντικά ακόμα από ό,τι στο παρελθόν. Το θέμα δεν είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής, είναι ένα θέμα στρατηγικής. Μιλάμε για το μεγάλο γεωστρατηγικό παιχνίδι τα επόμενα 50 χρόνια από σήμερα και αν δεν το αντιμετωπίσουμε σαν τέτοιο φοβάμαι ότι θα χάσουμε το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο αυξάνει την αλληλοεξάρτησή μας. Εμείς όμως στην ουσία εξαρτώμεθα όλο και περισσότερο. Δεν υπάρχει καμία μορφή αμοιβαιότητας από τις χώρες που έχουν πηγές αερίου και πετρελαίου και αυτή η εξάρτηση προσφέρεται για εκμετάλλευση. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Το βασικό συνεπώς πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι το ότι οι πηγές ε, βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες θα έλεγα είναι έφλεκτες και δεν μπορούμε εμείς να τις πάρουμε από εκεί η μόνη λύση είναι να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε τις περιοχές αυτές λιγότερο έφλεκτες και αυτή είναι η στρατηγική θα έλεγα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο τρόπος για να το πετύχουμε μπορεί να είναι μονομερής ή κοινός. Προς στιγμή θα έλεγα η μεμονωμένη αντίδραση κυριαρχεί αυτό φαίνεται από το ότι υπάρχει αντίσταση για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς στην Ευρώπη και κάποιοι από εμά εξακολουθούμε να είμαστε ε, θα έλεγα φυλακισμένοι ε, στις αλλαγές διάθεσης των Ρώσων και των Ουκρανών. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική εσωτερική αγορά. Η Ρωσία και αυτή παίζει το στρατηγικό της παιχνίδι, θέλει να επανατοποθετηθεί αμφισβητώντας το κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά από τον ψυχρό πόλεμο. Θέλει να ξαναγράψει τους κανόνες η Ρωσία και θέλει να βρεθεί σε καλύτερη θέση από αυτήν που βρίσκεται. Αυτό δεν το καταδικάσουμε γιατί αν ήμασταν Ρώσοι το ίδιο θα κάναμε αλλά θα πρέπει όμως να το αναλύσουμε αυτό σαν πρακτική και να δούμε ε, ποιες είναι οι καλύτερες μορφές αντίδρασης. Σχετικά με τον Αμπούκο θα ήθελα εδώ να τονίσω προς τον πρώτο ομιλητή ότι για την Ρουμανία εμείς από την αρχή θεωρήσαμε ότι το South Stream είναι ανταγωνιστής του Ναμπούκο το θέμα δεν είναι πόσα χρήματα μπορούμε να κερδίσουμε αν κάνουμε ε, το South Stream να περάσει από τα χωρικά μας ύδατα. Το θέμα είναι πολιτικοστρατηγικό. Το South Stream είναι ανταγωνιστής που θέλει να σκοτώσει τον Αμπούκο, τον καημένο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θα αμφισβητήσει επίσης και τις πηγές ε, του Ναμπούκο μέσω της δημιουργίας του South Stream και πείθοντας όλους τους συμμετέχοντες στο Ναμπούκο να πάνε ε, στο South Stream. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται στις χώρες οι οποίες υπογράφουν όχι μόνο το Ναμπούκο αλλά και το South Stream. Οι Ρώσοι δεν έχουν κανένα δισταγμό να ε, προκαλέσουν προβλήματα σε αυτούς οι οποίοι προσπάθησαν να βοηθήσουν τη Ρωσία και αυτό δείχνει ότι όταν πραγματικά περάσουμε στο ψαχνό η Ρωσία θα είναι στιγμή και δεν θα έχει κανένα δισταγμό να ακολουθήσει εγωιστικά εθνικιστικές τάσεις. Ο κύριος Ονισκίεβιτς αντιπρόεδρος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να εμβαθύνω λίγο αυτό που είπε ο Πάσκο. Να σας ρωτήσω γιατί καθυστερούμε με τον Αμπούκο Έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Υπάρχει αίσθηση ότι δεν συμβαίνει τίποτα για τον Ναμπούκο. Δυστυχώς οι πιθανοί προμηθευτές του Ναμπούκο στην ουσία προσελκύονται από τους Ρώσους να υπογράψουν ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με την Gazprom έτσι ώστε το φυσικό αέριο από το Αζερβαϊτζάν και το Καζακστάν να το στρέψουν στους ρωσικούς αγωγούς. Αυτό είναι κάτι που έχουμε πει στα ψηφίσματά μας, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εμπλακεί δίδοντας χρήματα, επενδύοντας χρήματα όπως το έκανε και στην περίπτωση του Γκαλιλαίου. Γιατί το Ναμπούκο έχει στρατηγική σημασία και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Το άλλο θέμα είναι το εξής. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε με την Ρωσία δεν είναι μόνο ότι η Gazprom είναι ο μονοπωλιακός παραγωγός αερίου, αλλά είναι και ο μοναδικός που μεταφέρει το αέριο, ελέγχει πλήρως ε, τους αγωγούς. Υπάρχει μία εξαίρεση, ένας αγωγός στη Ρωσία που δεν ανήκει στην Gazprom, το CPC, ο αγωγός της Κασπίας δηλαδή. Ο αγωγός αυτός ε, ελέγχεται από εταιρείες πετρελαϊκές όπως η Chevron. Δεν ελέγχεται μόνο από το ρωσικό κράτος ε, όπως η αγωγή της Gazprom. Και γι' αυτό λοιπόν αν πραγματικά έχουμε ένα τέτοιο αγωγό που περνάει από ρωσικό έδαφος αλλά δεν ελέγχεται από τους Ρώσους αυτό θα ήταν κάτι το θετικό το υγροποιημένο αέριο τώρα. Η τεχνολογία αναπτύσσεται. Νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για την εξαέρωση εκ νέου του υγροποιημένου αερίου. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε αν είναι ελκυστικός ο τρόπος χρήσης του υγροποιημένου για την νότια τουλάχιστον Ευρώπη. Ο κύριος Ρόφσιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας έχουν πει. Θα ήθελα να αναφέρω ένα πολύ μακροχρόνιο, αν θέλετε, και μακρόπνοο θέμα που έχει να κάνει με τον Βόρειο Πόλο. Λιώνουν οι πάγοι και ο Βόρειος Πόλος, η Ακτική Θάλασσα, σε μερικά χρόνια, σε πέντε χρόνια και λιγότερο, θα είναι ελεύθερη πάγου. Και φαίνεται ότι υπάρχουν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου κάτω από τον Βόρειο Πόλο και η Δανία της οποίας είναι αναπόσπαστο τμήμα η Γρυλανδία είναι αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία προσπάθειας ανάπτυξης αυτών των πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και αυτό θα μας οδηγήσει σε ε, υγροποιημένο αέριο το οποίο μπορεί να προκύπτει από αυτή την περιοχή. Μιλάμε για τεράστιους πόρους και φυσικά υπάρχει διελκυνστίνδα μεταξύ της Δανίας, του Καναδά και της Ρωσίας για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτών των κοιτασμάτων και η Δανία προσπαθεί να πείσει το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη να επιλύσει το πρόβλημα αυτό και ζητούμε και από τους ε, άλλους εμπλεκομένους να συμφωνήσουν μια τέτοια επιδίκαση αλλά αν θέλουμε να το δούμε αυτό μακροπρόθεσμα αυτό, αυτή μπορεί να είναι μια εναλλακτική ή μια πρόσθετη, μια παραπληρωματική πηγή ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος. Αν είχαμε πολύ καλές διασυνδέσεις του ενεργειακού δικτύου, του δικτύου ηλεκτροπαραγωγής, θα μπορούσαμε να είχαμε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλο και περισσότερο καθώς χρειαζόμαστε όλο και περισσότερη ε, ενέργεια αιωλικού χαρακτήρα, χρειαζόμαστε πολύ καλύτερες διασυνδέσεις του δικτύου αυτού. Θα, θα ζητήσουμε μία μελέτη για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τον Αρκτικό. Κύριος Κάλαμ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις ιδιαίτερα διαφωτιστικές πληροφορίες που μας έδωσαν. Αλλά νομίζω ότι τα συμπεράσματα αυτών των παρουσιάσεων είναι ότι η εποχή της παροχής φτηνού αερίου με ομαλή διαδικασία, με ομαλότητα παροχής, έχει ξεπεραστεί. Το φυσικό αέριο γίνεται όλο και πιο ακριβό και αυτό το οποίο μας σοκάρει είναι ότι τα προβλήματα του South Stream έχουν συνδεθεί με πολιτικά λάθη. Μερικές χώρες ελπίζουν ότι θα έχουν φτηνό φυσικό αέριο μέσα από εναλλακτικού αγωγούς φυσικού αερίου που προσφέρονται από τη ρωσική πλευρά. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο επόμενο χρονικό διάστημα γιατί θα υπάρξουν αυταρχικά καθεστώτα και δικτατορίες που δεν θα είναι τόσο αξιόπιστα και θα έχουν μεγαλύτερο πειρασμό που θα νιώθουν να χρησιμοποιήσουν σαν πολιτικό μοχλό το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Έρχομαι λοιπόν σε αυτά τα οποία είπε ο κ. Μόνακαν για την ανάγκη να ενισχύσουμε τη συνεργασία με ομονοούντες εταίρους. Να ενισχύσουμε λοιπόν τις διατλαντικές μας σχέσεις. Γιατί χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αξιοπιστία και μεγαλύτερη αλληλεγγύη, όπως τόνισε και ο συνάδελφος Πάσκο. Έχουμε ενώπιον μας τα δύο κέρατα του διλήμματος να κάνουμε μία προσέγγιση η οποία θα είναι ατομική και κοντόφελμη ή μια μακροχρόνια στρατηγικού χαρακτήρα. Να το πράξουμε αυτό όλοι μαζί. Δύο ερωτήματα τώρα για την αποδοτικότητα του πρωτοκόλου, των πρωτοκόλων της ενεργειακής χάρτας. Ξέρουμε ότι ο κ. Κόσετσε, ο Ρώσος πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, μας είχε πει πριν από ένα χρόνο περίπου ότι η Ρωσία υπέγραψε την ενεργειακή χάρτα όταν ήταν αδύναμη και καχεκτική. Τώρα όμως είναι έτοιμη να την επαναδιαπραγματευτεί. Γιατί έχει να κάνει με καταναλωτές και όχι παραγωγούς. Το άλλο ερώτημα είναι αν η Ρωσία μπορεί να παραγάγει αρκετό αέριο, γιατί οι στατιστικές δείχνουν ότι η παραγωγή της Gazprom τελματώθηκε τα τελευταία 8 χρόνια στο ίδιο επίπεδο. Και αυτό είναι και επίπεδο της πολιτικοποίησης αυτής της εταιρείας. Κύριε Σέβεριν, δεν θα επαναλάβω κύριε Πρόεδρε τα επιχειρήματα τα οποία έχουν αναφερθεί από τους διαφόρους συναδέλφους. I just want to make a short uh, note uh, saying that indeed uh, the resources are placed in volatile areas